Okay, ας ξεκινήσουμε, συνάδελφοι, γιατί έχουμε αυτή την κακή συνήθεια πάντοτε να ξεκινάμε καθυστερημένα ούτω ή άλλω εδώ στο Κοινοβούλιο. Πρωτού ξεκινήσουμε, θα ήθελα δύο υπενθυμίσει στου συναδέλφου να δώσω. Αύριο έχουμε μια κοινή ακρόαση με την Επιτροπή του Ντρουά, δηλαδή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε ό,τι αφορά την, ε, το συγκεκριμένο αν θέλετε, χώρο για την κοινωνία των πολιτών ε, στο PHS 5003 θα λάβει χώρα αυτή η συνεδρίαση. Σήμερα το πρωί εξετάσαμε και το ζήτημα ε, τη χρηστή διακυβέρνηση και τη σχετική έκθεση ε, που ασχολήθηκε και με το ζήτημα αυτό του συνεχνούμενου αν θέλετε, πεδίου δράση για την τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών και επίση στι 4 και 15 αύριο θα, υπάρχει μια κοινή ακρόαση για την Africa Rising, δηλαδή τον αυξανόμενο ρόλο της Αφρικής, γιατί βέβαια ουσιαστικά θα συζητήσουμε εκεί τις ε, συμφωνίες EPA και θα ακούσουμε και από την πλευρά των Αφρικανών εταίρων μας πώς τις αντιμετωπίζουν. Στο Γιάν 6Q2 αύριο στις 4 και 4 θα λάβει χώρα αυτή η ακρόαση. Ε, οπότε οι συντονιστές ε, θα μπορούσαν ενδεχομένω να υπενθυμίσουν εδώ στους υπόλοιπους ευρωβουλευτές. Το θα λάβουν χώρα αυτέ τι δύο ακροάσεις και να περάσουμε τώρα στο θέμα μας. Έχουμε και χαίρομαι πολύ έναν ε, υπουργό ε, από την πλευρά της Σλοβακίας, υφυπουργό ε, για τις εξωτερικές υποθέσεις και ευρωπαϊκές υποθέσεις της Σλοβακίας, που είναι αρμόδιος για αναπτυξιακά ζητήματα και άλλες επιτυχές σε αναπτυξιακής πολιτικής και ήδη γεμάτησε με τους συντονιστές, οπότε μας κοινοποίησε και κάποια από τα ζητήματα που θέλει να ασχοληθεί. Έχουμε και βέβαια τον ε, Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων τη Μάλτα, τον κύριο Τζορτζ Βέλα και τον καλωσορίζουμε θερμά, ε, γνωρίζουμε πώ ε, ήδη περιλαμβάνεται στην ομάδα συνεργασία με την Σλοβακή Προεδρία. Οπότε είναι πολύ καλό που είστε που συμμετέχει σε αυτέ τι συνεργασίε και για το γεγονό ότι είστε σήμερα εδώ μαζί με του συμβούλου σα, με του οποίου βέβαια και με εσά αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνεργασία, τη συνεργασία μα και ήδη τώρα στο πλαίσιο τη Σλοβακική Προεδρία. Ελπίζω λοιπόν πώ θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε μέσα στου ερχόμενου μήνε ε, στενά. Ο κύριο ε, Πάρισεκ θα ασχοληθεί κυρίω με ζητήματα ανθρωπιστική ε, βοηθεία. Υπάρχουν και πολλά ζητήματα τα οποία καλύπτει αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια και τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Είχαμε το Μάιο την Παγκόσμια <clears throat> Ανθρωπιστική Διάσκεψη στη Κωνσταντινούπολη και έχουμε και τον Ενρίκη ο οποίο είναι ο μόνιμος εισηγητή μα σε καταστήματα ανθρωπιστική ε, βοήθεια, ε, και ο οποίο ε, έχει εκπονήσει λοιπόν, και σχετική έκθεση από την δική μα πλευρά, οπότε θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων σε συνέχεια ακριβώ τη διαστήψη τη ανθρωπιστική διαστήψη κορυφή στην Κωνσταντινούπολη. Βέβαια, συνεχίζεται και η προσφυγική κρίση και συζητήσαμε χθε με τον Γενικό Διευθυντή τη ΔΕΦΚΟ σε ό,τι αφορά το Migration Compact, δηλαδή ένα είδο γέφυρα, αν θέλετε, μεταξύ διαχείριση του προσφυγικού αφενό και ανθρωπιστική βοήθεια εταίρου. Οπότε, να δώσω το λόγο σε εσά, ε, κύριε Υπουργέ, και μετά στου ε, συναδέλφου. Ευχαριστώ, Λίντα, αξιότιμα μέλη. Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι ενώπιόν σα για να συζητήσουμε τι προτεραιότητε τη Σλοβακική Προεδρία ε, στην ανθρωπιστική βοήθεια. Ορισμένοι διαπιστώσατε ότι σα κάναμε ένα μικρό δώρο ε, αυτά τα σημειωματάρια και το στήλο της Προεδρίας ελπίζω να είναι χρήσιμα. Ε, πραγματικά εκτιμούμε το έργο το δικό σας, της Επιτροπής σας, ειδικά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ανθρωπιστική βοήθεια. Πριν έρθω στην παρουσίαση του προγράμματός μας, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τους Ολλανδούς συναδέλφους και σας αξιότιμα μέλη για την ομαλή μετάβαση και αλλαγή της σκητάλης στην Προεδρία. Είναι πολύ ευχάριστο να παίρνει κανείς τη σκητάλη από τους Ολλανδούς, οι οποίοι πραγματικά είναι πολύ γνωστοί για την προσήλωσή τους. Όπως είπε η Υπουργός Μπλούμεν, ε, όταν ανέλαβε Κίνα, οι μεγάλες αλλαγές ε, χρειάζονται πολύ καιρό, άρα δεν μπορούμε όλα να τα ε, καλύψουμε στην εξάμηνη διάρκεια της Προεδρίας. Όπως είπατε και εσείς, θα εργαστούμε ως ομάδα και θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε τη δουλειά που έκανε η προηγούμενη Προεδρία. Και ο Υπουργό Εξωτερικών της Μάλτας που θα μας διαδεχτεί. Ε, είμαι βέβαιο ότι συμφωνεί. Επίσης όλοι συμφωνούμε ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στον κόσμο είναι πάρα πολύ δεινή. Την τελευταία δεκαετία η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοστάτησε και στην ε, ανθρωπιστική βοήθεια αλλά και σε νέα και πιο αποτελεσματικά μέσα κατά τη διάρκεια της ίδιας περίοδου όπως γνωρίζετε. Διπλασιάστηκε περίπου ο αριθμός των ανθρώπων που πλήττονται από ανθρωπιστικές κρίσεις. Στην Συρία και μόνο ο πόλεμος δημιούργησε τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Τώρα έχουμε μια κατάσταση όπου πάνω από 76 εκατομμύρια άνθρωποι από 31 χώρες χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι πάνω από 51 εκατομμύρια άνθρωποι που έχουν εκτοπιστεί λόγω πολέμου. Παραμένουν τέσσερι χώρε που θεωρούνται υψίστου επίπεδου προτεραιότητε και έκτακτη ανάγκη που είναι η Συρία, το Ιράκ, το Νότιο Σουδάν και η Εμένη. Βλέπετε πόσο διαφορετική είναι η κατάσταση σε σχέση με το έτος 2004 όταν η Σλοβακία άρχισε να δίνει ανθρωπιστική βοήθεια και να συμμετέχει σε αυτή τη συνεργασία και την ανθρωπιστική βοήθεια ως ε, νέο μέλος της Ένωσης το 2004. Ε, στην Κωνσταντινούπολη λοιπόν είχαμε πρόσφατα τη διάσκεψη ε, την παγκόσμια ε, για να έχουμε μέσα πιο ευέλικτα και πιο προβλέψιμα και πιο ικανά να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Παρά το γεγονό ότι αυξάνεται η συμμετοχή ε, των δωρητών, ε, είναι δύσκολο να ανταποκριθούμε στι αυξανόμενε ανάγκε. Ε, η ανθρωπιστική βοήθεια από μόνη τη, όσο σημαντική και να είναι, δεν μπορεί ούτε να αντιμετωπίσει ούτε να μειώσει καν σημαντικά τι αυξανόμενε ανάγκε εκείνων που έχουν ιδιαίτερα προβλήματα τώρα. Γι' αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το κακό στη ρίζα του που προκαλεί μαζικές ροές προσφύγων και εσωτερικά εντοπισμένων, να σταματήσει να τερματίζονται οι πόλεμοι, αυτό με ηγετική στάση των ηγετών μας και θα πρέπει να καλυφθεί και το έλλειμμα και το κενό ανάμεσα στην αναπτυξιακή βοήθεια και την ανθρωπιστική. Έχουμε ε, τρεις προτεραιότητες βασικές και τέσσερις ειδικέ. Ε, θα σας παρουσιάσω πρώτα τις βασικές. Η πρώτη είναι ε, βελτιωμένη και συντονισμένη απάντηση ανθρωπιστικής της κρίσης. Θα επικεντρωθούμε στο να βρούμε τρόπους να βελτιώσουμε την ανθρωπιστική μας ε, απόκριση με δράση συντονισμένη και συνεπή κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις τέσσερις χώρες που σας ανέφερα ε, και υπάρχουν και κάποιες συχασμένες κρίσεις που έχουν χαθεί από τα ραντάρ και θα πρέπει να ξανάρθουν στην ανθρωπιστική ατζέντα. Το προσφυγικό. Η Σλοβαγική ε, Προεδρία το θεωρεί προτεραιότητα, ε, καθώς επίσης και την αναγκαστικό εκτοπισμό και την ανθρωπιστική κατάσταση προσφύγων εσωτερικά εκτοπισμένων, καθώς επίσης και των κοινοτήτων και των κοινωνιών που τους υποδέχονται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να συνεργαζόμαστε με τους ανθρώπους επιτόπου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κατακαιρματίζεται η βοήθεια, θα πρέπει να είναι βιώσιμη και αυτό είναι το ε, πλεονέκτημα των αδράς τοπικά και λογοδοτούν και εκείνοι που παίρνουν τη βοήθεια. Ε, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο λοιπόν η τοπική κοινωνία και θα πρέπει αυτό να το αναγνωρίσουμε. Ε, Υπάρχουν τρόποι λοιπόν λειτουργία για να ανταποκριθούμε σε αυτά. Δεύτερο βασικό στοιχείο για μας και προτεραιότητα είναι να δώσουμε ε, συνέχεια στην Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης του Μαΐου. Πολλοί από εσάς συμμετείχαν εκεί. Η ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί σε πάνω από 600 στόχους για καλύτερη διεθνή και εθνική βοήθεια. Είχα την ε, τιμή να είμαι μέλος της αποστολής με τον πρόεδρό μου και θέλω να πω ότι πραγματικά είναι πολύ διάστατη η ε, προσέγγιση. Και να τονίσω τρεις διαστάσεις. Πρώτη, η πολιτική. Έχουμε συγκεντρώσει ε, παγκόσμια υποστήριξη από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα, αλλά και πρακτική επιτόπου ε, να δρούμε για να είναι περισσότερη και αποτελεσματικότερη η δράση μας και επίσης έχει και ένα χαρακτήρα συνειδητοποίησης, δηλαδή συγκέντρωσε την προσοχή της παγκόσμιας ε, κοινότητας η διάσκεψη ε, υποστηρίζει πολλές από τις μεταρρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είχε ζητήσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση και την εκπαίδευση. Επίσης, τόνισε αυτό που θεωρούμε και εμείς πρώτη μας προτεραιότητα. Η ανθρωπιστική βοήθεια δεν μπορεί να είναι ένα επαόριστον ε, υποκατάστατο πολιτικών λύσεων. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ε, τους πολέμους στη ρίζα τους και ε, τις ανθρωπιστικές κρίσεις παντού στον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεργαζόμαστε και με άλλους τομείς όπως είναι η ασφάλεια και η ανάπτυξη. Εδώ δεν έχει δοθεί συνένεση οριστική και μπορούμε να κάνουμε εμείς προσπάθεια κατά τη διάρκεια της Προεδρίας. Επίσης, ε, επίκειται και ε, η ε, Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και Σύνοδος Κορυφής των ηγετών μεταξύ κρατών μελών θα φροντίσουμε να βρούμε λύσεις βιώσιμες για τα προβλήματα της μετανάστευσης. Θα πρέπει να μιλούμε σαφώς και με μία φωνή στα διεθνή φόρα. Επιπλέον, θέλουμε να τονίσουμε την ανάγκη ε, να τηρείται το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, η ασφαλής πρόσβαση σε εμπόλεμες περιοχές και ε, βοήθεια καθώς επίσης και ιατρικό προσωπικό επιτόπου. Ε, το τόνισε και ο πρόεδρος μας στην Κωνσταντινούπολη. Είναι σημασία, έχει μεγάλη σημασία μάλλον να προστατεύονται εκείνοι που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια και η δουλειά τους και η ζωή τους. Τρεις μέρες μετά από το τραγικό θάνατο που βρήκε μια γιατρός μας η Βερόνικα Ρασκόβα που ε, δούλευε στο Νότιο Σουδάν και την πυροβόλησαν και τη σκότωσαν ε, όταν οδηγούσε ένα στενοφόρο και επέστρεφε, ε, μάλλον πήγαινε μια ετοιμόγενη γυναίκα στο νοσοκομείο. Ε, βεβαίως η σύνοδος κορυφής αυτή δεν είναι το τέλος, ίσα ίσα είναι η αρχή. Ε, θα πρέπει να έχουμε φιλοδοξίες και να βασιστούμε στην πολιτική συγκυρία που έχει τώρα δημιουργηθεί και πολύ γρήγορα να υλοποιήσουμε τις συλλογικέ μας υποχρεώσεις που αναλάβαμε. Και η Σλοβακία υποστηρίζει όλες τις βασικές δεσμεύσεις. Και όπως ανακοινώθηκε από το χρόνο θα διπλασιάσουμε την ανθρωπιστική μας βοήθεια και ε, θα ενθαρρύνουμε και ιδιώτες ε, να κάνουν εμπορικές δωρεές και χορηγίες. Ε, τρίτη προτεραιότητα είναι να προωθήσουμε την Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανθρωπιστική Βοήθεια, καθώς είναι ακρογωνιαίος λήθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών στον τομέα αυτού. Από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις υπόλοιπες χώρες ε, είμαστε τμήμα της Task Force για ε, την εφαρμογή του δεύτερου σχεδίου με αποτελεσματικότητα, με συντονισμό και με υποστήριξη όλων αυτών για τα οποία έχουμε δεσμευτεί. Αξιότιμα μέλη, όπως σας ανέφερα προηγουμένως, πέρα από αυτές τις τρεις βασικές προτεραιότητες, έχουμε και τέσσερις θεματικές προτεραιότητες, που είναι το φύλλο, η εκπαίδευση σε έκτακτες ε, περιστάσεις, ε, ανθρωπιστική, ε, σύνδεση μάλλον ανθρωπιστικής βοήθειας με την αναπτυξιακή, επισητιστική ασφάλεια και διατροφή. Υπάρχει και μία διάσταση φύλου στις κρίσεις που πλήττει ε, πιο σφοδρά η κάθε κρίση τις γυναίκες και τα κορίτσια. Όχι μόνο σε θανάτους, σε κοινωνική και οικονομική ανισότητα, αλλά και βία με βάση το φύλο. Ε, μαθαίνουμε ότι 60% ε, θανάτων των μητέρων που θα μπορούσαν να είχαν πρόληφθει γίνονται σε περιπτώσεις ανθρωπιστικής κρίσης. Επιπλέον, μία στις πέντε γυναίκες πρόσφυγες έχουν υποστεί σεξουαλική βία ή παρενόχληση. 70% ε, των γυναικών ε, κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Συρία έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση ή βία με βάση το φύλλο. Οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι οι πρώτες που τα πληρώνουν σε τέτοιες περιπτώσεις και είναι διαφυσβήτητη η συνεισφορά τους στην ανοικοδόμηση μιας χώρας μετά τον πόλεμο. Δεύτερη θεματική προτεραιότητα είναι να λάβουμε υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών και των ανηλίκων μετά από καταστροφές και πολέμους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση. Σήμερα ε, το 25% των παιδιών που είναι σε ηλικία να πηγαίνουν σχολείο, δηλαδή περίπου 500 εκατομμύρια, ζουν σε ε, περιοχές που γνωρίζουν κρίση. 75 εκατομμύρια δεν πηγαίνουν σχολείο ή έχουν κακής ποιότητας εκπαίδευση ή κινδυνεύουν να φύγουν τελείως από το σχολείο. Ταυτόχρονα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εκπαίδευση και η παιδεία είναι αυτό που χρειάζεται περισσότερο η κρίση. Γιατί ε, έτσι μειώνεται η έκθεση των παιδιών σε καταστροφές και αυξάνεται η αντίστασή τους. Η ε, Προεδρία μας θα δώσει ιδιαίτερο ρόλο και έμφαση στην ενίσχυση της παιδείας και της εκπαίδευσης σε ανθρωπιστικές ε, επιχειρήσεις. Καλωσορίζουμε και χαιρόμαστε πλήρως για την ε, απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αυξηθεί η χρηματοδότηση από το 2% στο 4% της ανθρωπιστικής βοήθειας για το σκοπό αυτό. Δεν μπορεί να περιμένει ε, η παιδεία. Την περασμένη εβδομάδα επισκέφθηκα ε, προσφύγων στο Λίβανο, ο οποίος Λίβανος φιλοξενεί περίπου 1,5 εκατομμύριο Σύρους πρόσφυγες και 500.000 Παλαιστινίους πρόσφυγες. Έχει κατακεφαλή το μεγαλύτερο ποσοστό, δηλαδή ένας στους τρεις που ζει στο Λίβανο είναι πρόσφυγας είναι μια κατάσταση που δεν μπορεί σχεδόν κανείς από μας να φανταστεί. Η κατάσταση με συγκίνησε πάρα πολύ αυτά που είδα εκεί. Είδα ανθρώπους να κάθονται στη σκόνη, στο χώμα, με ε, προσωρινή στέγη, παραπήγματα και δεν μπορούν να ζήσουν μια κανονική ζωή. Στην κοιλάδα Μπεκά, ε, ε, πήγαμε εκπροσώπους του ΟΗΕ και της ε, είπα της αρμοστίας και συζήτησα με μια οικογένεια με 7 παιδιά. Ο πατέρας είναι διαβητικός και η μητέρα είναι η μόνη που δουλεύει για την οικογένεια, για 9 άτομα. Ε, έχει υπομειστεί όλο το κόστος και βεβαίως είναι και μεγάλη δαπάνη η θεραπεία του διαβήτη. Άρα τα παιδιά δεν έχουν καμία δυνατότητα να πάνε σχολείο φυσικά και να μορφωθούν. Θα πρέπει ε, να αποτραπεί ο κίνδυνος του να μεγαλώνουμε μια χαμένη γενιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα. Αυτή η επίσκεψή με έπεισε και πάλι ότι η παιδεία θα πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα. Ιδιαίτερα ε, σε εκείνους που είναι αναγκαστικά εκτοπισμένοι, έχουν εξαναγκαστεί. Ε, και περισσότερε περιπτώσει δεν πρόκειται για μία γενιά, αλλά για δύο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα τη παιδεία και θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μα και είναι και εθνική μα προτεραιότητα. Φέτο ε, έγινε μια πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα συστήματα αυτά, για εκπαίδευση σε καταβλισμούς προσφύγων στη Συρία ή σε γειτονικέ χώρες, μεταξύ αυτών και ο Λίβανος. Ε, προς το σκοπό αυτό έχουμε δεσμεύσει μισό εκατομμύριο ευρώ. Επίσης έχουμε βάλει ένα ειδικό πρόγραμμα για υποτροφίες για φοιτητέ από τη Συρία. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το Λίβανο και τη Συρία. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε και τι γίνεται με την Κένια και άλλες χώρες της Αφρικής που υποδέχονται στο έδαφος τους πρόσφυγες. Η κατάσταση που βλέπουμε τώρα μπορεί ακόμα να επιδεινωθεί. Και λόγω της ε, τρομερής ε, ξηρασίας ε, στην ε, Αιθιοπία ε, τα τελευταία χρόνια, 15 χρόνια και 18 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια. Δεν υπάρχει μαγική λύση φυσικά ούτε πανάκια. Θα πρέπει κάθε φορά να ανταποκρινόμαστε στην εκάστοτε ανάγκη. Τρίτη μεγάλη λοιπόν ειδική προτεραιότητα είναι να προωθήσουμε μεγαλύτερη σύνδεση και να συσχετίσουμε περισσότερο την ανθρωπιστική βοήθεια με την αναπτυξιακή. Ο αναγκαστικό εκτοπισμός και η ανθρωπιστική κρίση χρειάζονται παρεμβάσει πέρα της έκτακτης ανθρωπιστικής βοήθειας που είναι προσωρινή. Χρειάζεται μια ολιστική αντιμετώπιση, ανθρωπιστική βοήθεια και αναπτυξιακή βοήθεια για να έχουμε πιο βιώσιμη προσέγγιση. Δηλαδή, αν δώσει κάποιο ένα ψάρι, όπω λέει η παλιά παροιμία, θα φάει μια μέρα. Αν το μάθει να ψαρεύει, ε, θα έχει να τρώει για όλη του τη ζωή. Η ε, Προεδρία μας θέλει πραγματικά να γεφυρώσει αυτό το χάσμα της ανθρωπιστικής με την αναπτυξιακή βοήθεια. Και τέλος, θέλουμε να δώσουμε έμφαση, όπως και στο παρελθόν, στην επιστημιστική ασφάλεια. Αυτό δεν χρειάζεται επεξήγηση εδώ, ιδιαίτερα στην Επιτροπή σα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοστατεί στην επιστημιστική βοήθεια και στη διατροφική βοήθεια στι πιο ευάλωτε περιοχέ, αλλά ακόμα 800 εκατομμύρια άνθρωποι υποσυτίζονταν το 2015. Και αυτό έχει να κάνει με ακραία καιρικά φαινόμενα όπως είναι το Ελνίνιο που μπορεί να ενταθούν και να γίνουν ακόμα πιο ακραία ως ε, απόρρια της κλιματικής αλλαγής. Αυτά θα πρέπει από κοινού να τα αντιμετωπίσουμε τη διεθνή κοινότητα με ένα συνολικό τρόπο, ε, ε, με επισητιστική ασφάλεια μέσω της ανάπτυξης, όπως γίνεται και με την ανθρωπιστική ανάπτυξη και βοήθεια. Και τέλος, κυρίες και κύριοι, βασικός στόχος και καθήκον και ευθύνη μας είναι να βελτιώσουμε περαιτέρω την ανθρωπιστική μας απόκριση. Οι κρίσεις γίνονται όλο και πιο οξύες, όλο και πιο επίγουσες, όλο και πιο αισθητέ στην Ευρώπη. Θα πρέπει η ανθρωπιστική βοήθεια να είναι όχι μόνο πιο αποτελεσματική, αλλά και πιο βιώσιμη. Θα τα ξαναπούμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας και περιμένω ε, τα σχόλιά σας και τις συστάσεις σας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας μας δώσατε μια καλή επισκόπηση των προτεραιοτήτων σας. Δεν αποκλίνουν και από πολλά από αυτά που λέγαμε εμείς εδώ και μήνες. Το μόνο ερώτημα που έχω τώρα, εγώ οι συνάδελφοι, αφορά την τεράστια επίση για ανθρωπιστική βοήθεια με τόσους ανθρώπους που μετακινούνται για λόγους ασφάλειας διατροφικής και λέγαμε χθε ότι είχαμε περικοπές στον περιπολογισμό και για την ανθρωπιστική βοήθεια αλλά και για άλλα χρήματα τα οποία αφορούν αυτές τις δράσεις. Βλέπουμε λοιπόν τα χρήματα έχουν αφαιρεθεί από γραμμές που αφορούν την διατροφική ασφάλεια για να πληρωθεί το τουρκικό σχέδιο. Οπότε δεν ξέρω τι άποψη έχουν και οι συνάδελφοι που παρακολουθούν τα θέματα του προπολογισμού προσεκτικά. Γκερέρο πρώτα, θα δώσω το λόγο στον Ερίκη Γκερέρο και μετά στους υπολείπους συναδέλφους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πάτσε, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την ε, παρουσία σας και για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων σας ως Σλοβακική Προεδρία. Νομίζω ότι είναι καλή είδηση ότι ο επόμενος υπεύθυνος θα είναι Μαλτέζος. Δηλαδή, εμείς θα πετούσαμε πάντα να υπάρχει μια συντονισμένη απάντηση από κοινού που θα εφαρμόζεται από διαδοχικές προεδρίες σε σχέση με τις ανθρωπιστικές ε, κρίσεις που δεν θα επαναλάβω, ξέρουμε ποιες είναι και που έχουν μεγαλύτερη σημασία και βάρος από ό,τι στο παρελθόν. Δυστυχώ θα αυξηθούν σε σημασία αυτές οι κρίσεις και δεν θα υποχωρήσουν. Δηλαδή οι σειράξεις που θα μπορούμε να λύσουμε τίνουν να μηδενιστούν και εμφανίζονται συνεχώς νέες και περισσότερες μαζί με άλλα φυσικά φαινόμενα όπως το Ελληνίνιο όπως αναφέρθηκε Όλα αυτά λοιπόν σκεγγραφούν ένα ορίζοντα ανθρωπιστικών αναγκών που αυξάνονται και θα αυξάνονται τα επόμενα χρόνια όπου θα προστίθενται οι πρόσφυγες, οι κλιματικοί λόγω θεομηνιών και σειράξεων. Πιστεύω ότι αυτό που μας παρουσιάσατε όπως είπε η Λίντα συμπίπτει κατά βάση με τις προτεραιότητες που προασπίζουμε εδώ στις, ε, στην Επιτροπή μας διάφορες πολιτικές ομάδες από κοινού τα τελευταία χρόνια. Είχαμε και τις προτεραιότητες που μεταφέραμε στην ε, Σύνοδο Κορυφής για τα ανθρωπιστικά ζητήματα στην Κωνσταντινούπολη παρόλο που η παρουσία μας δεν ήταν τόσο ισχυρή όσο θα επιθυμούσαμε. Πάντως Επί της ουσίας, οι προτεραιότητές μας κατά βάση συμπίπτουν ακόμα και λεπτομερώς με αυτές της Σλοβακικής Προεδρίας. Θα ήθελα να αναφέρω κάποιες από αυτές τις προτεραιότητες. Καταρχάς νομίζω ότι μία από τις άμεσες δράσεις σας θα είναι η εφαρμογή των συμβασικών συμφωνιών κατά την διάσκεψη της ε, Κωνσταντινούπολης. Εσείς είπατε ότι μαζί με τις χώρες μέλη και την Ένωση αναλάβατε γύρω στις 600 ε, δεσμεύσεις περίπου. περίπου. Σε όλους τους τομείς που εξέτασε η διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή να μην μείνει κανένας πίσω, ε, να αυξηθεί η χρηματοδότηση και να αναζητηθούν νέες πηγές χρηματοδότησης και νέοι δωρητές με φρέσκο χρήμα. Η πιο ενεργητική στάση στην ε, λύση διενέξεων και συγκρούσεων που υπάρχουν. Η προώθηση της εφαρμογής του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και αυτό που ονόμασε ο ΟΗΕ επένδυση στην ανθρωπιά. Έχουμε βέβαια και τις συνδιαλλαγές στα πλαίσια αυτών των συμβιβασμών. Και γι' αυτό ακριβώ θεωρώ ότι με τρόπο συντονισμένο η χωρισμένη και ένωση θα πρέπει να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει. Για να αποτελέσουμε και παράδειγμα παγκοσμίω και για να προσπαθήσουμε να οθήσουμε και τους υπόλοιπους που έχουν αναλάβει παρόμοιες δεσμεύσεις να τις στηρίσουν. Υπό την έννοια αυτή να σας πω ότι το Κοινοβούλιο ανέκαθεν ήταν υπέρ μιας συνολικής εποπτείας της εφαρμογής των δεσμεύσεων που ληφθήκαν στην Κωνσταντινούπολη. Βλέπουμε ότι όχι μόνο στην Ένωση αλλά παγκοσμίω. και με τη βοήθεια του ΟΗΕ γίνεται προσπάθεια για την εφαρμογή ενό παγκόσμιου συστήματος που θα προσπαθεί να εποπτεύσει το βαθμό εφαρμογής των δεσμεύσεων μας. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ένωση και κατά συνέπεια η Σλοβακική Προεδρία θα πρέπει να κάνει τα απαραίτητα σχετικά με αυτό. Αξίζει τον κόπο να τονίσουμε ότι το Κοινοβούλιο ήδη ζήτησε από την Κομισιόν να μας υποβάλει το δεύτερο σχέδιο δράσης για την Ευρωπαϊκή Συνένεση Ανθρωπιστικής Δράσης συμπεριλαμβανομένης και μίας αναθεώρησης αυτής της Ευρωπαϊκής Συνένεσης ώστε να προσαρμοστεί αυτή στα τωρινά χαρακτηριστικά των ανθρωπιστικών κρίσεων. Εσείς συγκρίνατε την τωρινή κατάσταση με αυτή του 2004 λέγοντας ότι υπερδιπλασιάστηκαν οι ανάγκες αλλά βεβαίως ανάγεται στο 96 αυτή, αυτός ο συμβασμός, αυτή η συνένεση. Εδώ και 20 χρόνια λοιπόν έχει αλλάξει πραγματικά δραματικά η κατάσταση οπότε θα πρέπει να μας απασχολήσει εδώ στην Επιτροπή μας αυτό. Γιατί μας έχει απασχολήσει επανειλημμένως η αναθεώρηση αυτή. Επίσης θα πρέπει να συζητήσουμε και την εφαρμογή της συνένεσης αυτής στα πλαίσια της γενικότερης στρατηγικής που η Ένωση και η Κομισιόν μόλις υιοθέτησαν τώρα μάλιστα τον Ιούνιο και που παρουσίασαν την περασμένη εβδομάδα στο Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο στην Ολομέλεια και που θα αναπτυχθεί περιττέρω στο Συμβούλιο, στις συζητήσεις κοινοβουλευτικές κλπ. Επ' αυτού να σας πω κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι αρκετά έτσι γενικευμένο στην Επιτροπή μας. Δηλαδή να προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε τις ιδιαιτερότητες της ανθρωπιστικής δράσης ως ίδιες. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι εμείς δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε την ανθρωπιστική βοήθεια σε σχέση με την ανάπτυξη και δεν πρέπει επίση να εθελοτυφλούμε για θέματα ασφάλεια τα οποία συνδέονται με την ανθρωπιστική βοήθεια. Θα θέλαμε όμω οι δράσει, οι αρχέ τη ανθρωπιστική βοήθεια, η ανεξαρτησία, η ιδιαιτερότητα, τόσο πάντων αυτέ οι βασικέ αρχέ, θα πρέπει να διαφυλαχτούν όταν θα πρέπει να εφαρμόσουμε μια προσέγγιση η οποία θα πρέπει να είναι καθαρά ασφάλειας ή από τη σκοπιά της ασφάλειας. Και τέλος, επειδή συμφωνούμε για τα θέματα φύλου και εκπαίδευσης, θα τα θίξουν και συνάδελφοι στη συνέχεια. Έχουμε πιέσει την Κομισιόν για τα θέματα φύλου και εκπαίδευσης ώστε να φτάσουμε στο 4% του συνόλου ανθρωπιστική βοήθεια. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν από την Προεδρία ω Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε και να πιέσουμε σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια ώστε να υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό όπως υπάρχει το 4% που σας αναφέρω προηγουμένως να υπάρχει ένα αντίστοιχο για την εκπαίδευση. Τέλος θα ήθελα να αναφερθώ στο ότι θα πρέπει να υπάρχει ομοφωνία μεταξύ μας και έτσι θα πρέπει να πάμε ομονοούντες στην ε, διάσκεψη του Σεπτέμβρη για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Να ρωτήσω λοιπόν, έχετε μήπως αρχίσει τη δουλειά για κάποιες προπαρασκευαστικές θέσεις του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της Ένωσης εν αυτής της διάσκεψης. Το είπε προηγουμένω, προηγουμένως. Βέβαια δεν θα μιλήσω για τις περικοπές και τα δημοσιονομικά όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια και τα θέματα της διατροφικής ασφαλείας και τη σχέση μεταξύ ανάπτυξης και διατροφής. Φαίνεται ότι αναβλήθηκε η διάσκεψη του Ρίου που έπρεπε να έχει γίνει το Σεπτέμβρη. Αλλά το θέμα αυτό ούτως ή άλλως θα πρέπει να το ξαναπιάσουμε με οποιοδήποτε τρόπο γιατί είναι απαραίτητο. Αυτά από μένα ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή τύχη. Ευχαριστώ Ανδρίκη. Αναζαμπόσκα. Γκέρεν, Ρόιμπουργκ, Χολβένι. Άρα υπάρχουν άλλοι που επιθυμούν το λόγο εκτός από αυτούς που ανέφερα. Όχι. Πολύ ωραία. Έχουμε χρόνο. Ζαμπόφσκα πρώτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μιλήσω σλοβακικά γιατί είναι σημαντική μέρα αυτή για την σλοβακική δημοκρατία. Καλώς ορίσατε λοιπόν κύριε Υπουργέ Εξωτερικών στην Επιτροπή μας, την Επιτροπή Ανάπτυξης. Είμαι εδώ στην Επιτροπή αυτή 13 χρόνια και με χαρά σας βρίσκω σήμερα. Από ό,τι είπατε για την ανθρωπιστική βοήθεια και το πρόγραμμα της Λογικής Προεδρίας συνεχίζεται στην ουσία το Ολλανδικό πρόγραμμα με τις για την παγκόσμια ανθρωπιστική διάσκεψη. Μου φαίνεται λοιπόν λογικό η Σλοβακία να προσπαθήσει να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί. Μία από τις φιλοδοξίες σας εδώ σε αυτό το τομέα είναι η βελτίωση του συστήματος παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως τα γνωρίζετε πριν λίγες μέρες, το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο αποφάσισε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια της Ένωσης στην Αφρική, στην περιοχή των μεγάλων λιμνών, κοστίζει υπερβολικά. Και σύμφωνα με το Ελεκτικό Συνέδριο, η Κομισιόν δεν διαθέτει επαρκείς πληροφορίες για να διερευνήσει κατά πόσο η βοήθεια αυτή είναι οικονομικά αποτελεσματική γιατί πάνω από το εμείς του προπολογισμού διοχετεύεται μέσω των υπηρεσιών των ΗΕ και δεν υπάρχει κάποιο feedback, κάποια αξιολόγηση αυτής της βοήθειας. Και είμαι βέβαιη ότι αυτό το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τις μεγάλες λίμνες, όπως συχνά συμβαίνει και με άλλα προγράμματα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω Προσπαθώντας να βελτιώσετε λοιπόν το σύστημα της ανθρωπιστικής βοήθειας θα αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό στο σύνολό του στο Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό θα πιέσετε την Κομισιόν να πετύχει περισσότερη διαφάνεια από τις υπηρεσίες του ΟΗΕ. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Παριζέκ για την εξαιρετική του παρουσίαση. Δεν έχω να πω τίποτα. Είναι καταπληκτικά, καταπληκτική παρουσίαση, θαυμάσια. Οι προτεραιότητε ταυτίζονται με τι δικές μας προσδοκίε. Ε, απομένει το ερώτημα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από κοινού. Είναι κοινό το εγχείρημά μα και θα πρέπει να προχωρήσουμε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει εκεί που υπάρχουν προβλήματα, όπως είναι η χρηματοδότηση και θα πρέπει να τα δούμε αυτά στο προσεχές μέλλον. Έχουμε και ένα θέμα συντονισμού της πολιτικής ανθρωπιστικής δράσης. Η δική μας επιτροπή πηγαίνει ακόμα παραπέρα. Εμείς έχουμε και την αναπτυξιακή βοήθεια στο χαρτοφυλάκιο. Εσείς είσαστε υπεύθυνοι για την επιβίωση εκείνων που βοηθούμε και εμείς είμαστε υπεύθυνοι και για τη διαβίωση εκείνων που επιβιώνουν. Έτσι να το πω με όρους κάπως απλοϊκούς. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν από κοινού. Νομίζω ότι έχουμε πραγματικά πολλή δουλειά μπροστά μας από κοινού. Το θέμα είναι πώς να διαφυλάξουμε την αμεροληψία ε, της ανθρωπιστικής βοήθειας στα πλαίσια της ε, συμφωνίας με την Τουρκία. Ο Επίτροπός μας που κάνει καταπληκτική δουλειά ε, δέχεται κατηγορίες που στιγματίζουν και δακτυλοδείχνουν αυτή την πολιτική γιατί θεωρείται ότι μεροληπτούμε στη συμφωνία με την Τουρκία, ε, της οποίας η πολιτική και ο πρόεδρος δεν είναι της αρισκείας όλων, για να το πω έτσι, μην πω τίποτα χειρότερο. Η ανθρωπιστική δράση, λοιπόν, δεν θα πρέπει να ε, γίνεται αντιληπτή ως, πώς να το πω τώρα, κάτι που συμφέρει ε, τις άλλες υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είμαστε στην υπηρεσία άλλων. Έχουμε εδώ ένα στεγανό, ένα σιλό, το οποίο εγώ θέλω να υπερασπιστώ. Ε, είναι κάτι ξεχωριστό. Ε, για να ανταποκρίνεται ε, στις έκτακτες ανάγκες και να μην πέφτει θύμα σε πολιτικά παζάρια ε, και χρειάζεται προσοχή και θα το προσέξουμε. Θα ήθελα λοιπόν να εισάγω και μια κοινοβουλευτική διάσταση. Εδώ εμείς, η Επιτροπή μας, είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο με τις κυβερνήσεις και χαιρόμαστε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Αλλά και εσείς από πλευρά σας θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια για το πώς σκέφτεστε να εμπλέξετε περισσότερο τα εθνικά κοινοβούλια σε αυτή την προσπάθεια και να υπάρχει εκεί ένα συντονισμός. Τελευταίο, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας θα μπορούσατε να μας ενημερώνετε για τις ανάγκες, τις συγκεκριμένες όμως ανάγκες που απαιτούν όλες οι θεομηνίες και τα δράματα και οι τραγωδίες που ανακύπτουν ε, κατά καιρού. Μπορεί να σας φαίνεται αυτό ευκαταφρόνητο ε, η λεπτομέρεια, αλλά δεν είναι εύκολο κάθε φορά να έχουμε τα στοιχεία. Μπορείτε να τηρείτε έτσι έναν κατάλογο μόνιμο, μια απογραφή των αναγκών. Αν μη τι άλλο για να το χρησιμοποιούμε στη συζήτηση για τον προπολογισμό. Σας ευχαριστώ και πάλι και μπορείτε να ε, προσβλέπετε και να υπολογίζετε στη δική μας ε, βοήθεια και υποστήριξη στα πλαίσια ε, της άσκησης των καθηκόντων σας. Ευχαριστώ. Κυρία Κυρία Χόιμπουκ, είστε λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ευχαριστώ, θέμα κύριε Πάζη, για την παρουσίασή σας στον όσο σκοπεύετε να κάνετε μέσα στο επόμενο εξάμεινο. Είπατε ότι θέλετε πως ε, ε, θέλετε να υπάρχει μια καλύτερη σύνδεση μεταξύ της ε, αναπτυξιακής βοήθειας και της ανθρωπιστικής βοήθειας, τους ώστε να έχουμε περισσότερα αποτελέσματα. Αναφερθήκατε στο παράδειγμα της εκπαίδευσης και πραγματικά είναι ιδιαίτερα εύστοχο αυτό το παράδειγμα, γιατί πολλοί από τους πρόσφυγες από τη Συρία επέστρεψαν γιατί ακριβώ ήθελαν να επιστρέψουν στα σχολεία του ε, τα παιδιά και δεν ήθελαν να υπάρξει μια χαμένη εντό εισαγωγικών ε, γενιά. Ε, και το ζήτημα τη αγορά εργασία προφανώ είναι ένα επίση εύστοχο ε, παράδειγμα, αλλά αναφέρθηκε επανειλημμένα βέβαια το πρόβλημα της ε, χρηματοδότησης. Ε, πέρυσι υπήρξε μια πολύ μεγάλη τρύπα στον προπολογισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας, οπότε θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η δική σας ιδέα, πώς θεωρείτε ότι θα μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε τέτοιου είδους δράσεις και να διασφαλίσουμε τα κονδύλια τη χρηματοδότηση. Ε, μεγάλοι φορη, σημαντική τη ανθρωπιστική βοήθεια, όπω η Ρωσία, δεν συμμετείχαν στη διάσκεψη κορυφή στην ε, Κωνσταντινούπολη. Οπότε σα ρωτώ πώ μπορούμε να εμπλέξουμε και πάλι τόσο σημαντικού φορεί σε αυτέ τι δράσει. Και ε, ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα να κάνω, το οποίο νομίζω πω αναφέρατε και εσεί στην παρουσίασή σα, ε, δηλαδή αυτό το ζήτημα των επιθέσεων κατά των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται στον ανθρωπιστικό τομέα. Εσεί αναφερθήκατε σε μια η οποία ε, σκοτώθηκε ο πυροβολισμό όταν οδηγούσε ένα στενοφόρο. Οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω τι μπορούμε να κάνουμε για να διαμορφώσουμε με πιο ασφαλή τρόπο, να καταστήσουμε πιο ασφαλή την εργασία των ανθρώπων οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να κάνουν αυτή την εργασία. Γιατί δεν είναι κάτι το αυτονόητο, δεν πηγαίνουν εκεί να βοηθήσουν ε, για να κερδίσουν περισσότερα χρήματα. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον ανθρωπιστικό από την πλευρά τη για να βοηθήσουν στην προστασία αυτών των ανθρώπων. Ευχαριστώ, Λεπρόεδρος. Ο κύριος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και να σας ε, συγχαρώ για το φιλόδοξο πρόγραμμα της ε, Προεδρίας σας. Ε, ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση που μας κάνατε γιατί έχετε ένα πολύ συγκεκριμένο και πολύ σαφές πρόγραμμα και μια δομή των όσων θέλετε να κάνετε και συμφωνώ πλήρω με τον συνάδελφο που αναφέρθηκε ότι ένα κέριο ζήτημα είναι η παιδεία. Και ε, επισκέφθηκα επανειλημμένα περιοχές της Συρία στο Ιράκ και στο Λίβανο και ε, διαπίστωσα ότι πραγματικά πρόκειται ένα από τα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Οπότε θα ήθελα ε, να μου πείτε τι ακριβώς θέλετε να κάνετε πιο συγκεκριμένα ω ε, ως αυτό το, project στον τομέα τη εκπαίδευση. Ε, και εδώ έχουμε δύο σημαντικά στοιχεία. Καταρχήν την εμπειρία των, τοπικών εθνών και στον τομέα τη ε, παιδεία. Ε, και βέβαια εδώ δεν θα πω ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε θέσει εργασία, ίσω είναι λίγο υπερβολικό, αλλά α δώσουμε τη δυνατότητα να λάβουν χώρα δράση σε τοπικό επίπεδο. Οπότε, ποια ε, είναι τα δύο κύρια, δύο κύριοι τρόποι για να παραμείνουν οι άνθρωποι στι ενεργοπεριοχέ. Και εδώ θα αναφερθώ και σε κάποια σχόλια που κάνετε κι εσείς. Αναφερθήκατε στις τοπικές δυνατότητες που υπάρχουν. Οι ικανότητε δηλαδή αυτών των ε, περιοχών, τις οποίες θα πρέπει να λάβουμε πιο σοβαρά υπόψη μας. Αυτές λοιπόν οι ικανότητες θα πρέπει να εφίστανται σε αυτές τις ε, περιοχές και ειδικότερα σε χώρες όπως η Συρία ή το Ιράκ είναι δύσκολο να μπορούμε να, να, λάβουμε υπόψη μας ε, και να ακούσουμε την, τις κατατόπους ε, εμπειρίες. Ε, δηλαδή όλοι επισκέπτονται κάποια κέντρα εκεί, τις πρωτεύουσες και μετά έρχονται με τις εμπειρίες τους, αλλά στο Ιράκ και στη Συρία παρατηρούμε το εξή φαινόμενο. ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τους ε, πρόσφυγες. Προφανώς ε, διάφοροι κεντρικοί φορείς και διεθνείς ε, οργανισμοί που έχουν να στήσουν εδώ ένα πολύ εκτεταμένο έργο και βέβαια εδώ υπογραμμίζω μια ακόμα φορά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος Αλλά από εκεί και μετά είναι ζήτημα όπου έχουμε χριστιανούς, ε, μουσουλμάνους, γιαζίδι και ούτω καθεξής. Και οι αντίστοιχες εκκλησίες έχουν να παίξουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της ε, ανθρωπιστικής βοήθειας. Αλλά η, το, το δικό μας ε, πλαίσιο δεν μας επιτρέπει να δεχτούμε τέτοια υποστήριξη. Δηλαδή με βάση το σημερινό μας πλαίσιο ως θρησκευτική οργάνωση κανείς δεν έχει άμεση πρόσβαση στην ε, χρηματοδοτική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το, το, το, το θέμα εδώ. Προφανώς υπάρχουν κάποιοι έμεσοι τρόποι μέσω συνεργασιών να ε, έχουν πρόσβαση σε αυτά τα κοντήλα. θα πρέπει τελικά να προσεγγίσουμε πιο άμεσα αυτές τις οργανώσεις. Δηλαδή όλες αυτές οι θρησκευτικοί ηγέτες και όλες αυτές οι δομές, γιατί τελικά δεν πρόκειται για θέμα πίστης, αν κανείς πιστεύει όχι, είναι αυτή η δομή των θρησκευτικών οργανώσεων που υπάρχει, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λάβει υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ένα τελευταίο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω είναι κάτι το οποίο αναφέρατε ε, στο τελευταίο κομμάτι της ομιλίας σας σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή. Και για την κλιματική αλλαγή πραγματικά το έχουμε μια πολύ ετερόκλητη εικόνα. Ο καθένας δηλαδή έχει να, να, να κάνει τις δικές του παρατηρήσεις και έχει τις δικές του σκέψεις. Νομίζω όμως θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο συνεκτικοί, να επικοινωνούμε και να έχουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια το τι θα πρέπει να συμβαίνει, για παράδειγμα, ποιος είναι, ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας ε, για ε, μια συγκεκριμένη περιοχή για τη μετακίνηση των ανθρώπων. Δεν είναι δηλαδή ε, κάτι το αφηρημένο όλο αυτό η κλιματική αλλαγή για τους εμπειρογνώμονες και για τις αναπτυγμένες χώρες. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και βέβαια ε, αντιλαμβάνομαι ότι δεν αφορά μόνο για μήκος τη μας Επιτροπή, αλλά θα ήθελα να δώσετε έμφαση πραγματικά ε, σε αυτό το ζήτημα και θα ήθελα ακούσω τελικά και κάτι, ότι θα, κάτι θα έχει γίνει στο τέλος της Πρόεδρας. σα. Νόης, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Λίντα. Και σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πάρτσακ, για την παρουσίασή σας και για την προετοιμασία σας ως προς το τι σκοπεύετε να κάνετε μέσα στο εξάμενο κατά το οποίο θα έχει η Σλοβακία την Προεδρία του Συμβουλίου. Ε, θα ήθελα βέβαια η χρονική συγκυρία να ήταν διαφορετική, δηλαδή να μην είχε μόλις συμβεί το Brexit, να μην βρισκόμαστε ενώπιον της προσφυγικής κρίση. αλλά τώρα βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση και έχετε πραγματικά πάρα πολλά ε, να κάνετε, πολλά θέματα να επιλύσετε, οπότε σας συγχαίρω για την πολύ καλά δομημένη ε, προετοιμασία σας. Σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η προηγούμενη Προεδρία, η Ολλανδική Προεδρία, μας υποσχέθηκε ότι θα ασχοληθεί επισταμένος και πολύ σοβαρά με τις υποχρεώσεις οι οποίες προέκυψαν από τη διάσκεψη της ε, Κωνσταντινούπολης. Οπότε θα ήθελα να σας δείσω και εσά. Ε, μέσα στο επόμενο εξάμεινο να εξετάσετε ποιο μπορεί να ανταποκριθεί στι υποχρεώσει του, ποιο ανταποκρίνεται στι υποχρεώσει του, έτσι ώστε τελικά να μπορέσουμε να ασκήσουμε και την σε επίπεδο ε, πιέσει, προκειμένου τελικά να φτάσει εκεί που πρέπει η ανθρωπιστική βοήθεια και να βελτιωθεί η συνεργασία και ο συντονισμό μεταξύ των χωρών. Ε, χαίρομαι για το γεγονό ότι αναφερθήκατε σε κάποιε κρίσει οι οποίε έχουν ξεχαστεί λίγο και στο γεγονός ότι αναφερθήκατε και στους εσωτερικά εκτοπιζόμενους, δηλαδή εντό της ίδιας χώρας, γιατί συχνά εμείς εξετάζουμε μόνο τους πρόσφυγες εκείνους οι οποίοι εγκαταλείπουν τη χώρα τους, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί πρόσφυγες μέσα στις ίδιες χώρες, εκτοπισμένοι μέσα στην ίδια χώρα. Και η προσέγγιση που υιοθετείται ότι δηλαδή θα πρέπει να υποστηρίξουμε τους πρόσφυγες και σε περιφερειακό επίπεδο, γιατί ακριβώ οι περισσότεροι πρόσφυγε θέλουν να παραμείνουν στην ίδια περιοχή, είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Ε, εμείς θα πρέπει να προσέξουμε και εδώ ειδικότερα στη δική μας Επιτροπή, έτσι ώστε οι νέες προσεγγίσεις που εθετούμε σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια και η συνεργασία με την ασφάλεια, θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ποιε εγγυήσει έχουμε σε ό,τι αφορά αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια, τι επιτυγχάνεται δηλαδή σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση τη ένδυση και ούτω καθεξή και ποιε είναι οι σχετικές, ε, τα σχετικά μέτρα ασφαλεία. Για παράδειγμα, μπορούν να υπάρξουν κάποιες αλληλεπικαλύψει σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, για παράδειγμα, αστυνομικών δυνάμεων, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποφύγουμε ότι ε, τα κλασικά εντό εισαγωγικών κονδύλια τη ανθρωπιστική βοήθεια να χρησιμοποιηθούν και κατά συνέπεια να είναι κατάχρηση των κονδυλίων για άλλου σκοπού. Σε ό,τι αφορά τώρα το στόχο του 4% για τον τομέα τη παιδεία, νομίζω πω είναι κάτι πολύ σημαντικό το οποίο θα μπορούσε να υποστηρίξει και η δική σας ε, Προεδρία. Σε ό,τι αφορά την αλληλεγγύη τώρα, μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πω ότι δεν κάναμε αρκετά για την ε, Ιταλία, την Ελλάδα και τη Μάλτα κατά τα πρώτα χρόνια, όταν άρχισαν δηλαδή να καταφθάνουν εκεί οι πρόσφυγες. Η κατάσταση έχει βελτιωθεί τότε αλλά ε, ακόμα δεν έχουμε φτάσει εκεί που θα έπρεπε σε ό,τι αφορά την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Και για να είμαι πολύ διπλωματικός να πω ότι η δική σα χώρα ε, σε ό,τι αφορά την πρόταση που έκανε η Επιτροπή για την Κατανομή των Προσφύγων δεν ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδης. Ε, οπότε θα ήθελα να ακούσω ε, από εσά πώ σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα. Γιατί θέλουμε να υπάρξει μια αλληλέγγυα κατανομή των προσφύγων, οπότε καλό θα ήταν η Προεδρία του Συμβουλίου δηλαδή η Σλοβακία αυτό το εξάμεινο, να δώσει το καλό παράδειγμα για να επιτύχουμε κάποια πρόοδο. Ε, δεν το αναφέρατε μέχρι τώρα, αλλά ξέρω από προηγούμενες συζητήσεις ε, θέλετε να εστιάσετε και στη βιώσιμη ανάπτυξη στις χώρες που λαμβάνουν ανθρωπιστική βοήθεια και αυτό είναι πραγματικά θετικό γιατί δεν ε, χρειάζεται μια ad hoc απόφαση που θα πρέπει να λεφθεί. Υπάρχει δηλαδή μια στοχοθέτηση που θα πρέπει να ερωτηθεί εδώ και στην Επιτροπή μας και στο Κοινοβούλιο ε, προς αυτή την κατεύθυνση με μεγάλο χρονικό ορίζοντα έτσι ώστε οι άνθρωποι γενικά στις περιφέρειες να έχουν πρόσβαση και στην ενέργεια. Ε, θα δώσετε βέβαια στα τέλη του 2016 τη σκητάλη στη Μάλτα και ε, μόλις έλαβε χώρα η κοινή ε, διάσταση μεταξύ χωρών και, και Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε φορά με εκνευρίζει το γεγονός όταν ε, κάθε κράτος μέλος ε, πρόκειται να αναλάμβει ε, την Προεδρία, όπως αυτή την περίπτωση η Μάλτα, δεν έχει τη διάθεση να φιλοξενήσει αυτήν την διασύψη μεταξύ χωρών και, και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε θα ήθελα να σας ζητήσω να πιέσετε την επερχόμενη Προεδρία που θα σας δεχτεί, δηλαδή της Μάλτας, να φιλοξενήσει αυτήν την ε, διάσκεψη, ούτως ώστε να δείξουμε και τη φιλοξενία μας απέναντι σε αυτές τις ε, χώρες. Έχετε πολύ φιλόδοξους στόχους, τους οποίους ε, θέσατε στον εαυτό σας και φαντάζομαι ότι στα τέλη του εξαμήνου σας θα μας αναφέρετε το τι έχετε επιτύχει και εάν επιτύχετε μόνο το 50% των όσων μας αναφέρατε σήμερα εδώ, θα έχει υπάρξει μια πραγματικά πολύ επιτυχημένη Προεδρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Νόρμπερτ. Ε, δεν νομίζω πως έχει ζητήσει κάποιο άλλο το λόγο, οπότε θα ήθελα να αναφερθώ μόνο σε κάτι που ανέφερε ο Νόρμπερτ σε ό,τι αφορά δηλαδή την, ε, ανθρωπιστική υπόδοχη δηλαδή, ε, και νομίζω πως αναφέρθηκε αυτό, δηλαδή το ζήτημα της κατανομής κάποιων κονδυλίων σε επίπεδο ανθρωπιστικής βοήθειας μεταξύ των ε, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει αναφερθεί αυτό ο τον δηλαδή ότι ήταν χειρότερη η κατάσταση στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, από ό,τι στις σειρές του Λίβανο. Οπότε θεωρώ πως ήταν πολύ θετική απόφαση που έλαβε η ΕΚΟ να αποδεσμευθούν κάποια κονδύλια από άλλες γραμμές του προπολισμού, ώστε να βελτιωθεί η ανθρωπιστική βοήθεια στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε ε, θα ήθελα να μα κρατήσει ενήμερου η Προεδρία ω προ το εάν βελτιώνονται τα πράγματα και η ΕΚΟ θα συνεχίσει να μα ενημερώνει και προφανώ ε, δεν ε, κατηγορούμε εμεί τι χώρε που υποδέχθηκαν του πρόσφυγες όπω την Ιταλία και την Ελλάδα αλλά πραγματικά θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σε θέση να υποδέχεται με τον κατάλληλο τρόπο αυτά τα, αυτούς τους πρόσφυγες και αναφέρομαι προφανώς ειδικότερα στις χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή μεταξύ αυτών και η Μάλτα. Ε, αφού έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που έχουν το πάντοτε υποχωρήσει που είναι φτωχότερες από τις δικές μας. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ όλους για τα υποστηρικτικά σας σχόλια για τις προτεραιότητες της Προεδρίας μας. Χαίρομαι που βρίσκουμε κοινό πεδίο συνεννόησης για αυτά και όπως είπε ο κ. αν πετύχουμε τα μισά θα είναι μεγάλη επιτυχία. Γι' αυτό ακριβώς Είπα στην αρχή ότι πρέπει να συνεχίσουμε από τους Ολλανδούς προκατόχους μας και να επιφέρουμε κάποια συνέχεια και να ακολουθήσουμε τα κοιμάλτα. για τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Έχω κάποια μηνύματα που μου έρχονται κατά νου επειδή συμφωνούμε όλοι ότι υπάρχει ανάγκη όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια για μια συνέχεια. Χρειάζεται καλύτερο συντονισμό και συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων ώστε αυτή η βοήθεια να είναι πιο αποτελεσματική. Επίσης, η αξιολόγηση και εφαρμογή των δεσμεύσεων της διάσκεψης αλλά και του θεματολογίου 2030. Νομίζω ότι αυτά πραγματικά είναι τα κυριότερα μηνύματα για τα οποία συμφωνούμε. Τώρα για τη χρηματοδότηση, Λίντα, όπως είπες και εσύ, ξέρουμε ότι η τωρινή κατάσταση επιδεινώνεται όσον αφορά τις ανάγκες. Συνεχώς. Πολλοί αριθμοί που ανέφερα προηγουμένως μας δείχνουν ότι υπάρχει μια ανθρωπιστική κρίση τεραστίων διαστάσεων το οποίο σημαίνει ότι αντιμετωπίζουμε πραγματικά τεράστιες προκλήσεις που επηρεάζουν κατά συνέπεια και τον προπολογισμό ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι το κάθε ευρώ θα δαπανάται αποτελεσματικά και θα πηγαίνει εκεί που πρέπει. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν είναι σημαντικό να αναφέρουμε και τη συμφωνία για την ανθρωπιστική βοήθεια και η χρηματοδότησή της θα πρέπει να γίνεται με τρόπο ευέλικτο και αποτελεσματικό και αυτό είναι ένα από τα κύρια συμπεράσματα της διάσκεψης. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε αυτή τη θαυμάσια δουλειά που ξεκίνησε με τις προηγούμενες προεδρίες και να την φέρουμε σπέρα Για το follow-up τώρα τη παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψης. Είναι αλήθεια ότι είχαμε μια αρκετά δύσκολη προπασκευαστική διαδικασία το καλοκαίρι με διαφορετικέ προσδοκίες. Συμμετείχαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, αλλά στο τέλο νομίζω ότι είχαμε καλή συμμετοχή της νους κυβερνήσεων, ΜΚΟ κλπ και καταφέραμε να βάλουμε στο προσκήνιο τα ανθρωπιστικά ζητήματα. Θα πρέπει λοιπόν τώρα να κάνουμε κι άλλα σε σχέση με το ανθρωπιστικό δίκαιο και την αποτροπή των σειράξεων, όπου όντως όλοι συμφωνούμε ότι εκεί θα πρέπει να συμμετάσχουμε πολιτικά, να έχουμε πολιτική παρουσία. Τώρα, για τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε, να δούμε πώς θα μπορούσαμε να τις εντονίσουμε και να εφαρμόσουμε κατά διάρκεια της Προεδρίας μας και να βρούμε και τον να δυνατό τρόπο εποπτείας τους. Και αυτός ο μηχανισμός εποπτείας μετά από τη μεγάλη συμφωνία που ανέφερα, ή σε συνδυασμό με τη μεγάλη συμφωνία που ανέφερα προηγουμένως. Επίσης, μιλήσατε για τη σχέση μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και ανάπτυξης προσωπικά θεωρώ ότι αυτό είναι από τα πιο ενδιαφέροντα ζητήματα των προτεραιοτήτων μας, γιατί πρέπει να πω ότι οι παραταμένες, οι εκτοπισμοί σήμερα δείχνουν μετά από 70 χρόνια εκτοπισμών ότι δεν μπορεί κανείς να βασίζεται μόνο στην ανθρωπιστική βοήθεια. Γι' αυτό ακριβώ είναι κεφαλαιόδου σημασίας κάποιος να μπορεί να ανοίξει μια κοινωνία και να, έχει, και να ζει μια αξιοπρεπή ζωή. Και αυτός είναι ο κυριότερος λόγος, ίσως για τον οποίο θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπαθίες μας και να δούμε πώς θα μπορούσαμε να συντονιστούμε με τρόπο αποτελεσματικό. Δηλαδή χρειάζονται πιο συνεκτικά προγράμματα ανάπτυξης με πολιτική δέσμευση, τηρώντας και σεβόμενοι βέβαια τις ανθρωπιστικές αρχές. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Συνένεση που λέγαμε για την ανθρωπιστική βοήθεια. Η συνένεση από μόνη της είναι εξίσου σημαντική σήμερα όπως ήταν το 2007. Μαζί με τους υπόλοιπους λοιπόν εταίρους μας θα προσπαθήσουμε να διαδραματίσουμε ένα ενεργό ρόλο για να συγκροτήσουμε ομάδες που θα εξετάσουν ακριβώς το πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά. Χαιρετίζουμε το γεγονό ότι το σχέδιο επικεντρώνεται και στοχεύει στα κυριότερα, δηλαδή ανθρωπιστικό δίκαιο, ανάγκες που υπάρχουν και πώς θα μπορούσαν να εφαρμοστούν όλα αυτά σε πρώτη φάση. Η κυρία Ζαμπόρσκα, η συναδελφός μου από τη Σλοβακία. αναφερθήκατε στην έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Χαιρετίζουμε την έκθεση αυτή. για την ομάδα εργασίας ΚΟΑΦΑ και θα δούμε κατά πόσο θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα του Συμφουλίου υπό τη δικιά μας Προεδρία η έκθεση αυτή. Και συγγνώμη που δεν σας στα Σλοβακικά, λέει ο Πρόεδρος τι άλλο, συντονισμός για τα οικονομικά το κάλυψα, χρηματοδότηση εκπαίδευσης, τι άλλο, τι άλλο. Αν είναι πολλοί από εσά αναφερθήκατε στην εκπαίδευση. και την σχετική προστασία των εργαζομένων στο ανθρωπιστικό κλάδο. Η εκπαίδευση δεν αφορά μόνο την παιδεία, αλλά το γεγονό ότι η εκπαίδευση και οι υποδομέ εκπαίδευση, σχολεία κτλ. πρέπει να αποτελούν ένα ασφαλή λιμένα. ώστε να μην στρατολογούν, ας πούμε, παραστρατικές ομάδες μαθητές ή να μην τους καταναγκάζουν σε υποχρεωτική εργασία από μικρή ηλικία ή τα κορίτσια να είναι αντικείμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Όλα αυτά θα είναι πολύ πιο δύσκολο να, να συμβούν αν τα παιδιά αυτά πηγαίνουν στο σχολείο και είναι κομμάτι μιας κοινότητας που εκπαιδεύεται. Θα πρέπει λοιπόν στα πλαίσια της εφαρμογής του ανθρωπιστικού δικαίου να κάνουμε τα σχολεία και τους τόπους εκπαίδευσης ένα ασφαλή λιμένα για αυτά τα άτομα. Οπότε έτσι εμεί αντιλαμβανόμαστε την εκπαίδευση, ένα στοιχείο που αποτελεί δηλαδή σημείο ασφάλειας τώρα για τους εργαζόμενους νομίζω ότι το κυριότερο εδώ είναι η εφαρμογή του ανθρωπιστικού δικαίου θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε όπου μπορούμε τα θεμελιώδη δίκαια ιδιαίτερα σε περιοχές σύραξης. Και τα τελευταία χρόνια είδαμε ότι παραβιάζονται πολύ συχνά αυτές οι μορφές δικαίου και έχουμε πολλά θύματα εργαζομένων που εργάζονται δηλαδή στον τομέα της παροχής βοήθειας. Οπωσδήποτε θα πρέπει να καλύψουμε και αυτό το θέμα και μεγάλη σημασία. Τώρα, το πώς θα μπορούσαν να εμπλακούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι στον τομέα αυτό ώστε να συμμετάσχουν στην διάσκεψη. Νομίζω ένα θέμα που αφορά την παγκόσμια κοινότητα αυτό. Αναφερθήκατε και στη Ρωσία. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας θα προσπαθήσουμε να εμπλέξουμε και τη Ρωσία και τους άλλους εταίρους μας στο πλαίσιο του ΙΕ και της Γενέβης. Θα έχουμε οπότε διασκέψεις και διασκέψεις κορυφής που θα γίνουν για τα θέματα αυτά και για την Ένωση βέβαια ως πρωταγωνιστή στα ανθρωπιστικά θα είναι σημαντικό να συμμετάσχουν και άλλοι σημαντικοί παράγοντες της ανθρωπιστικής βοήθειας. Όπως λέγαμε πριν, Πρέπει να έχουμε συμμετοχή και συντονισμό. Πρέπει να συμμετάσχουν όλοι. Γιατί υπάρχει έλλειψη κονδυλίων και πιθανώς η χρηματοδότηση να μην αρκέσει ποτέ. Πρέπει λοιπόν όλοι να συμμετάσχουν γιατί όλοι αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή όλοι έχουμε τον κοινό στόχο την επίλυση των ανθρωπιστικών κρίσεων. Αυτά τι άλλο, για να δω τι άλλο με ρωτήσατε. πώς να αποφύγουμε τις μετακινήσεις. Να μην δηλαδή οι κάτοικοι στον τόπο τους. Αυτό είναι εξίσου σημαντικό ζήτημα. Το είδαμε στο Λίβανο όταν συζητήσαμε με κυβερνητικούς αξιωματούχους και με εργαζόμενους. Θεωρούν ότι η διεθνής κοινότητα και ο ΙΕ και η ΕΕ δεν καταλαβαίνουν ακριβώς το πλαίσιο ή το τι ισχύει τέλος πάντων στο Λίβανο από τη στιγμή που το εντρίο του πληθυσμού είναι πρόσφυγες. Οπότε συμφωνώ με την εμπλοκή και τη συμμετοχή των τοπικών αρχών στην εφαρμογή όλων αυτών των προσπαθειών. Αυτό είναι μεγάλη σημασία γιατί οι τοπικές κοινωνίες πρέπει οπωσδήποτε να συμμετάσχουν και να εμπλακούν σε αυτές τις διαδικασίες γιατί πολλές φορές ε, έχουν αμφιβολίες σε σχέση με την ε, βοήθεια που διοικητεύεται προς τους πρόσφυγες τη στιγμή που μεγάλα κομμάτια του λιβανέζικου πληθυσμού βρίσκονται στο όριο της φτώχειας. Νομίζω ότι θα εκτιμούσαν οι Λιβανέζοι αλλά και αλλού αυτό μια επαφή μαζί τους, μια συνεργασία πριν την παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Νομίζω ότι τα κάλυψα όλα, όλα τα σχόλια, της παρατηρήσεις σας. Αν όχι, πολύ ευχαρίστως να τα πούμε και από κοντά. Έχω εδώ και την ομάδα μου που θα με εκπροσωπεί Θα έρχομαι πάντως να σας βλέπω και νομίζω ότι μπορούμε από κοινό να κάνουμε πολλά. Πάντως σημαντικό είναι να πούμε ότι όλοι είμαστε ακριβώς στην ίδια μοίρα, δηλαδή Κοινοβούλιο, Συμβουλίο, Κομισιόν, γιατί όσες πληροφορίες μοιραζόμαστε και ενημερώνουμε ένα τον άλλον, τόσο πιο εύκολο θα είναι βεβαίω να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι προκλήσει. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, Υπουργέ. Δεν βλέπω κανέναν να ανέβει και να λέει ότι δεν καλύψατε την ερώτησή του. Τα υπερκαλύψατε. Σας θυμίζω, συναδέλφοι, ότι στι 5 έχουμε κοινή ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για το θέμα του αναγκαστικού εκτοπισμού, ε, της αναγκαστικής εκτόπισης και θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε εκεί στις 5 η ώρα, όχι σε αυτή την αίθουσα, ούτε καν σε αυτό το κτίριο, αλλά στο Γιάν 2Q2. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της δουλειάς μας και κάνουμε και κοινή έκθεση με την Επιτροπή Εξωτερικών, όπως γνωρίζετε, γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Υπουργέ, θα τα ξαναπούμε. Με χαρά να συνεργαστούμε. Ξέρετε, το καλοκαίρι δεν θα έχουμε, ελπίζω, καμιά μείζωνα νέα ανθρωπιστική κρίση να ηρεμήσουμε λίγο, ε, γιατί τα έχουμε δει τα περασμένα καλοκαίρια, φεύγαμε για διακοπές και ξεσπούσαν φρίκες και τρομακτικά πράγματα καλοκαιριάτικα. Λοιπόν, ε, ε, ευχαριστήσουμε τον Υπουργό που μας ήρθε. Στο καλό. Okay, colleagues, if those who are leaving can leave. Λοιπόν, όσοι θέλετε να αποχωρήσετε, παρακαλώ, εσύ. Um, Πάμε λοιπόν στο σημείο 17 τώρα, το οποίο είναι ε, συζήτηση με θέμα τη Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης ΣΟΕΣ μεταξύ των κρατών της κοινότητας Ανατολικής Αφρικής. Παρακαλώ συνάδελφοι, αν θέλετε αποχωρήστε ήρεμα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα τώρα που θα συζητήσουμε για τις ΣΟΕΣ με τις χώρες ε, της κοινότητας Ανατολικής Αφρικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει αυτή τη συμφωνία, να δώσει τη συνένεσή τους. Πέντε είναι οι χώρες. Μπουρούντι, όπου ξέρετε τα προβλήματα, Κένια, Ρουάντα, Ταζανία και Ουγγάντα. Έχει απολύτω δίκιο ο εισηγητή ο κύριο ε, Πρέντα. Γίνεται τρομερή φασαρία. Θα αρχίσω τώρα να σα κατονομάζω. Και αφορά και την ίδια μα τη γραμματεία που κάνουν πηγαδάκια εδώ πέρα. Ησυχία για να μπορέσει ο κύριο Πρίντα να μα παρουσιάσει την έκθεσή του. Νομίζω είναι καλέ οι συνθήκε. πάρα πολύ σημαντική έκθεση κύριε Πρέντα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που παρέμειναν σήμερα στη συνεδρίαση en fait... Όντως, έχετε μια γνωμοδότηση στα χέρια σας. Είναι γνωμοδότηση, επαναλαμβάνω, επί της ουσίας είναι αρμόδια Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Η γνωμοδότηση αυτή ε, συνετάχθη με βάση τις μεγάλες κατευθυντήριες γραμμές ε, που είχαμε στις 20 Ιουνίου, πριν από λίγες μέρες. Και γι' αυτό το λόγο εγώ δεν θα επαναλάβω όλα τα σημεία που ήδη συζητήσαμε. Στις 20 Ιουνίου θα περιοριστώ στην παρουσίαση των συμπερασμάτων μου μετά από εξέταση του κειμένου συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κοινότητας της Ανατολικής Αφρικής. Γενικά νομίζω ότι αυτή η ΣΟΕΣ, EPA στα αγγλικά, θα δράσει ως καταλήτης για την ε, ανάπτυξη, βιώσιμη ανάπτυξη ενώ και χωρίς αποκλεισμούς στην περιφέρεια αυτή του κόσμου. Σε ό,τι αφορά τα αμυγός εμπορικά ζητήματα, επειδή είναι ασύμμετρη προς την αγορά η συμφωνία αυτή και επειδή επιτρέπει ε, στους εταίρους μας να εξαιρούν τους ευαίσθητους τομείς από την απελευθέρωση. Η συμφωνία αυτή διαφυλάσσει τα περιθωρία ελιγμών των χωρών εταίρων μας. Και εμείς επιμείναμε πάρα πολύ σε αυτό, να έχουν αυτή τη διακριτική ευχέρεια. Θυμίζω επίσης τις μακροχρόνιες ε, μεταβατικές περιόδους, μέχρι και 25 χρόνια, για ορισμένες κατηγορίες ε, προϊόντων. Επίσης, εξαιρέσεις από την ε, διάνοιξη των αγορών, ε, εγγυήσεις για τις αναδυόμενες ε, βιομηχανίες, την επιστημιστική ασφάλεια, την επιβολή εξαγωγικών φόρων και δασμών. Όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα δούμε σε μια συνολική προοπτική υπέρ της ανάπτυξης, γιατί αυτό μας διέπει στη λειτουργία αυτής της Επιτροπής. Επίσης, υπάρχουν κάποιοι κανόνες που διευκολύνουν τις ε, εξαγωγές και ε, τονώνουν την ε, περιφερειακή ολοκλήρωση που είναι βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια της σύναψης αυτών των συμφωνιών. Τώρα μπορεί να εκφράζουμε τη λύπη μας που δεν γίνεται σαφής αναφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη αυτό θα μπορέσει να επαναεξεταστεί μια πενταετία μετά τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας, ε, χάρη στην ε, αντίστοιχη ρήτρα. Μια επιτροπή υψηλών αξιωματούχων παρακολουθεί αυτή την υπόθεση, καθώς επίσης και τις επιπτώσεις που έχει στη βιώσιμη ανάπτυξη. Και πάντα από τη σκοπιά της ανάπτυξης αναφέρω ένα ουσιαστικό κεφάλαιο για την αναπτυξιακή συνεργασία, καθώς επίσης και ε, ε, θέματα που αναφέρονται στο παράρτημα και είναι θετικά γιατί αντανακλούν και τις ανάγκες αλλά και τα συμφέροντα των εταίρων μας καθώς επίσης και τις προτεραιότητές τους. Πλην όμως, όπως και για τις υπόλοιπες ΣΟΕΣ, το θέμα της χρηματοδότησης θα είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Ε, και θα πρέπει και εμείς βεβαίως να έχουμε ε, γνώμη, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να φροντίσουμε η εφαρμογή τους ε, να έχει τη δέουσα χρηματοδότηση, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές δυνατότητες απορρόφησης. Ανθρώπινα δικαιώματα και διακυβέρνηση γίνεται ρητή αναφορά στη χρηστή διακυβέρνηση και χαίρομαι γι' αυτό ε, μεταξύ ε, άλλων. Αν και θα ήταν προτιμότερο να είχαμε μια ρήτρα αυτόνομη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προς το παρόν θα πρέπει να ε, επαναπαυθούμε σε αυτό και να μας ικανοποιήσει το κεκτημένο της Συμφωνίας Κοτονού και γίνεται αναφορά σε αυτό. εκπνέει η Συμφωνία Κοτονού και μπορεί να είναι μια καλή αφορμή για ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει και εδώ να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να ζητήσουμε να ενισχυθούν οι ρήτρε ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο σύστημα μετά το Κοτονού. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, διότι πρόκειται να ψηφίσουμε την έκθεση του κυρίου Νόιζερ μετά το καλοκαίρι. Θα πω δύο λόγια για το μηχανισμό παρακολούθησης της συμφωνίας. Το είχαμε ξαναπεί και θε, τέλη Ιουνίου είναι μεικτή επιτροπή, όχι κοινοβουλευτική, συμμετέχει και η κοινωνία των πολιτών. Θα πρέπει να φροντίσουμε μετά τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας να υπάρχει ένας ισχυρός μηχανισμός παρακολούθησης και ε, πολύ συγκεκριμένα να υλοποιείται η συμφωνία και ξεκάθαρα. Και χαιρετίζω την προθυμία της κυρίας Μάλστρομ της Επιτρόπου να ασχοληθεί με αυτό το θέμα και το ανέφερε μάλιστα και σε επιστολή της που έστειλε την περασμένη εβδομάδα ε, στον πρόεδρο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, ίντα, συμπεραίνοντας. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι, ότι αυτή η συμφωνία εταιρικής οικονομικές σχέσεις είναι αρχή και μόνο. Τα πάντα θα εξαρτηθούν από την υλοποίηση και θα κρυθούμε εκ του αποτελέσματος. Η Επιτροπή μας θα πρέπει να έχει κομβικό ρόλο στην εφαρμογή της συμφωνίας αυτής. Και μια ερώτηση έχω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν μου το επιτρέπετε. Τι γίνεται με την υπογραφή της συμφωνίας αυτής, πότε θα γίνει, τον Ιούλιο, όπως είχε προβλεφθεί ή μήπως θα αναβληθεί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you very much. very clear report. Ευχαριστούμε. Ήταν πολύ σαφής ε, αυτή η παρουσίαση και πολύ οι συστάσεις που κάνετε και στην ε, έκθεσή σας. Ε, ο Νόμπαντ Νόζα έχει ζητήσει παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Λίντα και ευχαριστώ και τον Κριστιαν για την τοποθέτησή του. επί της αρχής δεν μπορώ να υποστηρίξω αυτό που υπόθηκε η τελευταία ε, συζήτηση, δηλαδή το Μπουρούντι, η Ουγγάντα, η Τανζανία, η Κένια ε, και οι υπόλοιπε χώρε που καλύπτονται ε, είναι οικονομικά σωστά ολοκληρωμένες, οπότε νομίζω πως θα πρέπει να προβούμε σε αυτή την προσφορά απέναντί τους ενιαία δηλαδή της μείωσης των σχετικών δασμών. από την άλλη πλευρά βέβαια μας λυπεί το γεγονός ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα περιβαλλοντικά ε, πρότυπα δεν ε, αναφέρονται ρητά. Υπάρχει απλά μια έμεση αναφορά στη Συμφωνία Κοτονού. Ε, πέραν των, ε, του σημαντικού πολιτικού ε, ζητήματος, ότι δηλαδή έχουμε ε, πάντοτε πει ότι σε όλες τις εμπορικές ε, συμφωνίες θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα ανθρωπιστικά, ανθρωπιστικά δηλαδή ανθρώπινα δικαιώματα, συγγνώμη, περιβαλλοντικά ζητήματα κ.ο.κ. ούτω τίθεται πέραν αυτού και το ερώτημα τι συμβαίνει πέραν τη συμφωνίες κοντονού. Για μας είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει μια σωστή εποπτεία της εφαρμογής στην πράξη των συμφωνιών EPA, έτσι ώστε να εντοπίζουμε ε, από νωρί ε, προβλήματα και να επιλύουμε προβλήματα που μπορούν να προκύψουν στις ε, χώρες της Ανατολικής Αφρικής και γι' αυτό είναι πολύ καλό το γεγονό ότι προβλέπεται η σύσταση μια συμβουλευτική επιτροπή ενό consultative committee. Επίση για μα είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει ενεργή συμμετοχή της Οργανωμένης Κοινωνίας των Πολιτών, ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στο Μπουρούντι. Ε, ήδη αναφέρθηκα στην ανάγκη δηλαδή περαιτέρω διαλόγου για ανθρώπινα δικαιώματα. Όμως από χθε το βράδυ έχουμε νέες εξελίξεις γιατί η ε, μελέτη για την οποία είχε δώσει εντολή ε, στο Κέμπριτς ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει λοιπόν δημοσιευθεί και η εν λόγω λοιπόν έκθεση φτάνει στο συμπέρασμα ότι αυτές οι EPA οι οποίες ε, συνάπτονται με τις χώρες της Αφρικής ε, δεν μπορούν στο πλαίσιο του μηχανισμού συντονισμού του κοτόνου να θεωρηθούν ως κατάλληλα μέτρα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, οι εμπειρογνώμονες μας λένε εδώ ότι οι συμφωνίες τις οποίες συνάπνουμε με τις χώρες της Ανατολικής Αφρικής αναφέρονται ναι μεν ε, στην ανθρωπιστική ρήτρα, αλλά εδώ, σε αυτές τις τελευταίες συμφωνίες, η Επιτροπή έχει επιλέξει διαφορετική διατύπωση στις εν συμφωνίες. Άρα, κατά τη δική μας άποψη θα πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω αυτό το ζήτημα γιατί γνωρίζω ότι ε, ακόμα και στη δική μου ε, πολιτική ομάδα υπάρχουν ισχυρές αντιστάσεις απέναντι στην σύναψη τέτοιων συμφωνιών εάν δεν επιληθεί αρχικά το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δηλαδή τι ακριβώ θα συμβαίνει στο επίπεδο των συμφωνιών σε περίπτωση παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δηλαδή, ε, στι συμφωνίε τι αντίστοιχε ε, ε, με το Καριφόρου, με την Νότια Αφρική, με τη Δυτική Αφρική, τα πράγματα είναι διαφορετικά από τι συμφωνίε με την Ανατολική Αφρική. Οπότε θα πρέπει επιτέλου η Επιτροπή να μα δώσει κάποιε εξηγήσει. Γιατί ακολούθησε μια διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τις χώρες της Ανατολικής Αφρικής σε σύγκριση με τις άλλες τρεις περιοχές που ανέφερα μόλις τώρα οπότε θα ήθελα να μας δοθεί και ο κατάλληλος ε, τρόπος να παραταθούν λίγο οι σχετικές προθεσμίες για την υποβολή τροπολογιών και για την ψήφιση ούτως ώστε να λάβουμε αυτή την ενημέρωση που ζητάμε από την πλευρά της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Χόιμπουκ, παρακαλώ. Ναι, δεν πρόκειται εδώ για την πρώτη συμφωνία εταιρική σχέση την οποία συζητούμε και νομίζω πω είναι γνωστό από την πλευρά των ε, Πρασίνων εμεί υιοθετούμε μια μάλλον επικριτική στάση, ειδικότερα σε ό,τι αφορά αυτέ τι συμφωνίε με τι ε, χώρε τη Ανατολική Αφρική. Έχουμε δηλαδή ε, πέντε χώρες, ε, από τις πέντε χώρες τέσσερις ε, ανήκουν στις λιγότερο αναπτυγμένες και η Κένια είναι πιο αναπτυγμένη και ανήκει σε ένα διαφορετικό επίπεδο αν θέλετε οικονομικής ανάπτυξης. Από εκεί και μετά έχουμε την κατάσταση όπου η Τανζανία ε, αποφάσισε να μην προβεί στην υπογραφή αντίστοιχου συμφώνου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, αναφέροντα ω αιτία το Brexit. Και βέβαια κάτι τέτοιο θα έχει και περαιτέρω αρνητικό αντίκτυπο στην περιοχή. Δηλαδή θα έχει ε, αρνητικό αντίκτυπο καταρχήν στην Κένια, γιατί η Κένια ειδικότερα ε, χρειάζεται την πρόσβαση στην αγορά, χρειάζεται κατά συνέπεια μια τέτοια συμφωνία. Αντιθέτω, οι, υπόλοιπε ε, χώρε δεν θίγονται τόσο πολύ, ακριβώ γιατί ούτω ή άλλω δεν είναι τόσο οικονομικά αναπτυγμένε για να χρειάζονται αυτή την πρόσβαση. Οπότε, είναι προβληματικό το να περιλαμβάνουμε στην ίδια συμφωνία διαφορετικές χώρες με διαφορετικά συμφέροντα και διαφορετικό επίπεδο οικονομική ανάπτυξης. Δεν πρέπει να υιοθετούμε λοιπόν μια τέτοια ίδια προσέγγιση απέναντι σε χώρε με τόσο διαφορετικά προφίλ. Από εκεί και μετά αυτέ οι συμφωνίε ε, δεν ε, δημιουργούν κίνητρα για την διαφοροποίηση ε, της οικονομίας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή εξάγονται κυρίως τρόφιμα, οπρολαχανικά και μιλάμε για το 60% εδώ συνόλου των ε, εξαγωγών και είναι ενδιαθοκομείας, οπότε αφού μιλάμε ε, για ήδη ε, ελάχιστα ανεπτυγμένε χώρε, ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο τι πιέζουμε ακόμα περισσότερο προ τα cash crops και κατά συνέπεια δεν του επιτρέπουμε να δημιουργήσουν μια βιώσιμη, αυτόνομη οικονομία. Ουσιαστικά του ε, πιέζουμε προ την κατεύθυνση του να παράγουν για εξαγωγέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν νομίζω πω μια τέτοια προσέγγιση είναι σωστή. Μετά σε ό,τι αφορά την ε, πρόσβαση στην ε, αγορά, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη αυτή είναι περιορισμένη ακριβώς γιατί υπάρχουν και υψηλά επίπεδα προτύπων σε ό,τι αφορά την υγιεινή, δηλαδή υπάρχουν πολύ ψηλότερε απαιτήσει ε, και κατά συνέπεια η επεξεργασία των τροφίμων ε, γίνεται ακόμα πιο δύσκολη ακριβώς γιατί πρέπει να ε, τηρούνται σχετικά πρότυπα. Κατά συνέπεια το ζητούμενο είναι να ενισχύσουμε τις τοπικές εκεί αγορές και όχι να κατευθύνουμε την παραγωγή προς μια αγορά στην οποία ούτως ή άλλως δεν είναι έτοιμοι να έχουν πρόσβαση. Μετά αναφέρθηκα σε κάτι άλλο σήμερα στο οποίο στην ακρόαση και αυτό είναι τα διαφυγόντα έσοδα των κρατών στο επίπεδο της φορολογίας. Η προσέγγιση που μας ανέφερε σήμερα το πρωί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Collect More, Spend Better, αλλά να μείνουμε μόνο στο Collect More, ε, με, με τα EPA ουσιαστικά είμαστε πιο αυστηροί σε, σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις που ε, ε, ε, προβλέπουμε με βάση τα όσα προβλέπει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός ε, Παγκόσμιο Εμπορίου. Δηλαδή, ε, εμείς προβλέπουμε υψηλότερα τέλα, αλλά ενώ είπαμε ότι θέλουμε να έχουμε ε, αντίστοιχη μείωση των σχετικών ε, επιβαρύνσεων. Από την άλλη πλευρά βέβαια βρισκόμαστε σε τελείως διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης, οπότε για αυτές τις χώρες δυσκολεύουν πάρα πολύ τα πράγματα, ακόμα και αν υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις, να βρεθούν ακριβώς ναι, σε μια κατάσταση ισότιμης, αν θέλετε, μεταχείριση μεταξύ των χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των ίδιων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις διατάξεις ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ήδη σε αυτό αναφέρθηκε ο συνάδελφος Νόρμπαντ, ε, εδώ βέβαια σε αυτά συγκαταλέγονται και άλλε στόχοι όπω η βιώσιμη ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντο και τα σχετικά πρότυπα. Όλα αυτά λοιπόν, όλες οι πτυχές δεν περιλαμβάνονται παρκώ μέσα στι συμφωνίε EPA. Ε, και επίση. η ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών δεν είναι, ε, είναι επαρκώς ε, ε, για παράδειγμα αν θα ισχύουν τα πρότυπα ΕΛΟ, η περιβαλλοντικά πρότυπα ή ό,τι άλλο. Ε, Άρα λοιπόν αυτό που εγώ θα ήθελα να προτείνω είναι όχι να εστιάζουμε πάρα πολύ στην απελευθέρωση της αγοράς θα πρέπει να ε, ε, προωθήσουμε την ανάπτυξη των ίδιων των αγορών αυτών των χωρών και στο επίπεδο των περιφερειακών των χωρών τη Αφρικής, προτού τις κατευθύνουμε περισσότερο προς την ευρωπαϊκή αγορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Θα υπάρξει μια παρουσίαση όπως ανέφερε ο κ. Συνόσα αύριο στις 3 κοινή παρουσίαση στην Επιτροπή. Είναι σε σχέση με μια ε, έκθεση σε ό,τι αφορά τις σχετικές διατάξεις της συμφωνίας ε, EPA σε σχέση με τη συμφωνία Ε, Στον κύριο Πρέντα να πω ότι ναι, θα πρέπει να θέσουμε ένα ερώτημα στην Επιτροπή σε ό,τι αφορά την ε, Τανζανία. Γιατί αυτό που ακούμε είναι ότι δεν προτίθεται πλέον να υπογράψει τη Συμφωνία Τανζανία λόγω του Brexit. Θα θέλαμε να ακούσουμε κάτι από την Επιτροπή. Δηλαδή ότι από τη μία ακούμε ότι υπογράφει τη συμφωνία, από την άλλη η Τανζανία δεν υπογράφει λόγω Brexit. Και μετά, αυτό που ζήτησε ο κύριο Νόσο, δηλαδή η προθεσμία για την υποβολή τροπολογινών είναι αύριο. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν είναι επίγουσα αυτή η διαδικασία. Η Επιτροπή δηλαδή δεν έχει θέσει κάποιο, κάποια προθεσμία για την υποβολή το που λέμε μέχρι στιγμή, Οπότε ενδεχομένως θα μπορούσαμε να δώσουμε ε, στους συναδέλφου αν συμφωνείτε, όπως το κύριο Μέσο και άλλους, ε, τη δυνατότητα να υποβάλουν τροπολογίε, να τους δώσουμε μεγαλύτερη προθεσμία για να δουν ποιε είναι οι εξελίξεις. Αυτή τη στιγμή η προθεσμία είναι για αύριο το μεσημέρι για την υποβολή Ε, αλλά ε, παρότι θα βρούμε σε, σε ψηφοφορία, δεν έχουμε λάβει ακόμα το σχετικό αίτημα από το Συμβούλιο. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, α ακούσουμε πρώτα τι έχει να μα πει η Επιτροπή και μετά να αποφασίσουμε τελικά αν χρειάζεται να ψηφίσουμε ή αν καλύτερα να περιμένουμε μετά το καλοκαίρι να έχουμε περισσότερε πληροφορίε και μετά να ψηφίσουμε. Ο λόγο στην Επιτροπή. Εκτό μικρόφωνο. Κύριο Βάλ, λοιπόν, από τη Γενική Yes, dealing with economic ναι, για τι ε, συμφωνίε εταιρικών σχέσεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Μπρέντα για τη δουλειά που έκανε για αυτές τις συμφωνίες. και για την ε, καλή συνεργασία που είχαμε σε σχέση με αυτές τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Να αναφερθώ όμως σε, που, σε αυτό που είπατε εσείς, Πρόεδρε, το ότι χρειάζεται η Τανζανία περισσότερο χρόνο για την υπογραφή αυτής της συμφωνίας. Πρέπει να είμαστε βέβαια προσεκτικοί με τις διατυπώσεις μας. Δεν νομίζω ότι αποφάσισαν να μην υπογράψουν, τουλάχιστον δεν μας είπαν κάτι τέτοιο, οι άλλοι στην περιοχή. Ο λόγος αναβολής δεν είναι αυτός που φαίνεται. Ήρθα με καθυστέρηση και ζητώ συγγνώμη γιατί ήμουν δίπλα σε συνάντηση με τους περισβευτές των χωρών αυτών της Αφρικής και άκουσα τι είχαν να μας πούν και μας διαβεβαίωσαν ότι το θέμα της αναβολής είναι ένα θέμα ίσων σημασίας. Το οποίο και της Ένα απλό θέμα, όπως είπε και ο Ουγγανέζος, σα συγγνώμη. Και το μόνο που θέλουν είναι λίγο χρόνο παραπάνω να συμφωνήσουν όλοι να υπογράψουν ταυτόχρονα. Εμείς ανέκαθεν τους υποστηρίζαμε και τους αφήναμε χρόνο. Ποτέ πάντως δεν μας είπαν ότι το πραγματικό ζήτημα ουσίας εδώ για την υπογραφή ήταν το επανομαζόμενο Brexit. Συνεχίζουμε λοιπόν τη δουλειά μας από την Κομισιόν για την υπογραφή και επικύρωση από τις πέντε χώρες. Όπως είπαν και οι υπερσβευτές είναι οι πιο ενωμένοι περιοχή της Αφρικής αυτή. Θέλουν να προχωρήσουν μαζί. Θέλουν να πετύχουν τους στόχους ολοκλήρωσης που έχουν θέσει. Και όπως και εμείς ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα αποτελέσματα της συμφωνίας. Σημαίνω εδώ ότι η επιστολή της είναι κάτι το ευπρόσδεκτο, το χαιρέτησαν αποτελεί βάση εργασίας ώστε να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή και τον αντίκτυπο αυτής της συμφωνίας. Έχουμε και μία θεσμική δομή για να το κάνουμε αυτό, πάνω στην οποία βασιζόμαστε, σε υπουργικό αλλά και άλλα επίπεδα, επίπεδο κοινωνίας πολιτών, μέσω μιας συμβουλευτικής επιτροπής. και αν μου επιτρέψετε δεν θα αναφερθώ και τόσο στο ερώτημα του καθηγητού Βάρτ που από ό,τι καταλαβαίνω θα συζητήσουμε αύριο στην Κοινή Επιτροπή. Βεβαίως θα συζητήσουμε περισσότερο αλλά μπορώ από τώρα να σας απαντήσω το γιατί υπάρχει διαφορετική διατύπωση αυτές τις ρήτρε στη συμφωνία. Είναι επειδή διαπραγματευτήκαμε διαφορετικούς εταίρους που έχουν διαφορετικές ευαισθησίες. Το πνεύμα όμως υπό το οποίο διαπραγματεύτηκαν αυτές οι διατάξεις είναι ταυτόσιμο και εμπίπτει στο πνεύμα της Συμφωνίας Κοτονού και αύριο πάντως θα ρυθμιστούν αυτά τα θέματα και θα συζητήσετε αν θέλετε λεπτομέρειες με καθηγητή Μπάρτος. Και αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι ακόμα σχετικά με κάτι το οποίο δεν ήταν σαφές στο παρελθόν. για την μείωση της διαφοροποίησης των εξαγών από αυτή την περιοχή της Αφρικής μετά από τις συμφωνίες. Αυτό θεωρούμε δεν είναι ακριβές, είναι ανακριβές. Επειδή θεωρούμε ότι οι πιο ευέλικτοι κανόνες ακριβώς αποτελούν μεγαλύτερη ευκαιρία, ευκαιρία για εξαγωγές συγκεκριμένων προϊόντων προς την Ευρώπη. Απόλυ εισοδήματος τώρα, Πρόεδρε. Κάναμε τη δική μας ανάλυση που ευχαριστώ να σας μεταβάσουμε όταν ολοκληρωθεί, που δείχνει ότι η προσπάθεια φιλελευθερωποίησης στην περιοχή αποτελεί τη χαμηλότερη στην Αφρική για τον απλό λόγο ότι το 65% εισαγωγών από την Ευρώπη ήδη σήμερα βρίσκονται στο επίπεδο 0. Οπότε είναι λογικό να δείχνει η μελέτη ότι έχουμε πολύ μικρό αντίκτυπο, δηλαδή πολύ μικρή απολύτω οδήματος. για το άνοιγμα τώρα των αγορών υπό τις συμφωνίες αυτές. Αυτό, αν το πούμε, παραβλέπει το γεγονός ότι ε, μιλάμε για ποσοστά σε διάρκεια 25 ή 35 ετών από τις χώρες αυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστηρίξει αυτές τις χώρες ώστε να μπορούν από μόνες να αντιμετωπίσουν αυτές τις ε, προκλήσεις και η κυρία Γκαριμπάλντι, η παρακαθήμενή μου, αν χρειαστεί θα σας δώσει και τις απαραίτητες λεπτομέρειες σχετικά. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκαριμπάλντι από την ε, Γενική Δευκό. έτσι δεν είναι. Ναι, καλησπέρα. Ναι. Υπάρχει δέσμευση όσον αφορά την ανάπτυξη για συνεργασία σε διάφορους τομείς ώστε να ενισχύσουμε την εφαρμογή της συμφωνίας από την ΕΕ δεσμευτήκαμε για την χρήση οικονομικών και μη οικονομικών πόρων από τα εργαλεία μας εργαλεία που αφορούν βοήθεια για την ανάπτυξη και άλλα εργαλεία ώστε να αντιμετωπίσουν αυτές οι χώρες αυτό που θεωρούν πρόκληση σχετικά με την εφαρμογή. Αυτό βεβαίω θα πρέπει να συνοδεύεται ή μάλλον να συνοδεύει μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να αναλάβει η κυβέρνηση Χρειάζονται λοιπόν νομοθετικές μεταρρυθμίσεις όσον αφορά το επιχειρήν που πρέπει να συνεργάζονται επίσης και από φορολογικές μεταρρυθμίσεις κλπ. Επίσης συζητάμε με τις πέντε κυβερνήσεις τα σχέδια εφαρμογή, δηλαδή τα εθνικά σχέδια εφαρμογής, δηλαδή τα εθνικά σχέδια, όπου αναλύουμε κάποια ζητήματα μαζί με τις κυβερνήσεις, εξετάζουμε την εθνική κατάσταση, την κατάσταση σε κάθε χώρα και αναφέρουμε κάτι ως επικοινωνία, τη μορφή δηλαδή επικοινωνίας με τα διάφορα υπουργεία ή τις άλλες αρχές που σχετίζονται άμεσα με, τις, ε, με την εφαρμογή αυτών των συμφωνιών εταιρικής σχέσης στα πλαίσια της Κοτονού. Μαζί λοιπόν θέλουμε να εντοπίσουμε τα μέτρα που θα μπορούσαν να υιοθετήσουν οι κυβερνήσεις, πώς εμείς μπορούμε να τις βοηθήσουμε, ποιοι είναι οι τομείς που μπορούμε να βοηθήσουμε, ποιες είναι οι αλλαγές που θέλαμε να γίνουν ώστε να τους διευκολύνουμε να αυξήσουν τις εξαγωγές τους στην Ένωση. Αυτά λοιπόν τα σχέδια βρίσκονται σε προκατακτική φάση. Έχουμε ξεκινήσει διαβουλεύσει με τις κυβερνήσεις και θέλουμε να αρχίσουν αυτές τι διαβουλεύσεις αφού υπογραφούν οι συμφωνίες. Αυτό θα είναι και το κύριο κανάλι χρηματοδότησης. Χρηματοδότηση που προέρχεται από τα εθνικά και περιφερειακά προγράμματα και στοχεύει χρηματοδότηση σε κλάδους κλειδί, ενέργεια, μεταφορές, γεωργία, για τη διευκόλυνση του εμπορίου, κυρίως σε παραγωγικούς τομείς που προωθούν την παραγωγικότητα στις χώρες αυτές και τις βοηθούν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Να σταματήσω εδώ γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Έχουμε και άλλο ένα θέμα και πρέπει να τελειώνουμε σε λίγο. Αλλά εδώ είμαι, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι εδώ. Κύριε Πρέντα, ακούσατε και τους συναδέλφους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το μόνο που μπορείτε να αλλάξετε είναι να πείτε ναι ή όχι. Εμείς ε, ε ως κοινοβούλιο. Δεν ξέρω, πείτε μου πώ το βλέπετε. ε, τώρα εγώ τι να σα πω. Θα πρέπει να το αναβάλουμε, ε, σαφέ δεν είναι. Παρόλο που όσοι θέλουν να το απορρίψουν έχουν ε, κάθε διάθεση και όρεξη ήδη. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, τυπικά θα πρέπει να το αναβάλουμε και να περιμένουμε διευκρινήσεις για αυτά που ακούσαμε. Τώρα τι να σας πω εγώ. Απάντω ναι σε αυτό το αίτημα αναβολής. Σε ευθετότερη ημερομηνία δεν είναι έτσι δεν είναι. Ε, για πότε δηλαδή. Ε, να μην το πάμε Χριστούγεννα γιατί έχουμε και δουλειές. Ναι, έχετε και ο κόσμος θα ψηφίσει ναι ή όχι, αλλά θα πρέπει... Δεν μας ζήτησε το Συμβούλιο επίσημα να δώσουμε τη συγκατάθεσή μας. Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε τον Αύγουστο χωρίς να μας ρωτήσουν. 31 Αυγούστου συνεδριάζουμε, μπορεί μέχρι τότε μας έχουν ερωτήσει. Δεν έχει τροπολογίες, ναι ή είναι. Λοιπόν, θα ε, τα ξαναπούμε τέλη Αυγούστου και θα ορίσουμε και ημερομηνία. Δεν έχουμε άλλα θέματα. Ε, θα έχουμε αποφασίσει αν θα μπει μέσα ή έξω η Τανζανία κτλ. έχουμε τίποτα άλλο να προσθέσουμε, όχι. Ευχαριστώ πολύ, αλλά έχουμε άλλο θέμα εμείς, 18. Ερώτηση της κυρίας Χάουταλα για τη χρήση των κονδυλίων των αναπτυξιακών δεν θα σας διαβάσω όλη την ερώτηση. Να τα πει η Χάιντι καλύτερα. Σε ένα λεπτό όμως. Ευχαριστώ πολύ. Λίντα. Ποιο είναι το ζήτημα. Πρόσφατα παρατηρείται μια τάση που είναι εύκολο να τη δει κανείς. Έχουμε διάφορα αιτήματα από πλευράς κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπα τι εκπρόσωπο ζητάει και καμιά φορά και η να γίνονται μεταφορές πιστώσεων που είχαν σαφώς ε, μπει στην άκρη για την καταπολέμηση της φτώχειας και για στόχους αναπτυξιακής πολιτικής. Για αλότριους σκοπούς ε, είναι ε, υποτιθέμενη σύνδεση της ασφάλειας με την αναπτυξιακή βοήθεια. Και αυτό που με ανισχύει εμένα και με έχει θορυβήσει και άλλους είναι ότι δίνουμε και υποδομές στο στρατό των ε, χωρών εταίρων ε, για ανεπτυξιακή βοήθεια. Χωρίς να εκριζώνουμε τις πραγματικές αιτίες της φτώχειας. Έχει έρθει η ώρα να μας δώσει μια ε, απάντηση της προκοπής η Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ. Πώς το καλό εξηγείται αυτές τις αλλαγές. Ο κάθε πικραμένος έρχεται και παίρνει τα δικά μας λεφτά. Okay, thank you very much. Um, Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τον Κλάο Σκούτεσάλτε που είναι αναπληρωτής διευθυντής στην ΤΕΦΚΟ. Απλή ερώτηση, πώς σας φαίνεται. Ε, ε, δεν πιστεύω να έχει περίπλοκη απάντηση. Ο Κλάος έχετε το λόγο. Um, I will try to... Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να δώσω μια απλή απάντηση σε μια περίπλοκη ερώτηση, διότι είναι πολύ περίπλοκη ερώτηση ε, σε ό,τι αφορά τώρα το background. Αξίζει να θυμίσουμε ότι ως φορείς της ανάπτυξης όλο και περισσότερο εργαζόμαστε σε καταστάσεις κρίσης, πολέμων, ε, εύθραυστες ε, και είμαστε οι πρώτοι που έχουμε στο μυαλό μας. Αυτό το έχει πει και ο Επίτροπος ο ίδιος, αν δεν μπορούμε να έχουμε καταστάσεις που είναι κάπως σταθερές, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Δεν μπορούμε να αναπτύξουμε τις δικές μας προσπάθειες για την αναπτυξιακή βοήθεια. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένα αυτά τα δύο. Γι' αυτό και προτείναμε όλη αυτή τη δέσμη στις 7 Ιουλίου. Ένα ολόκληρο πακέτο εγγράφων είναι η ανακοίνωση για το πλαίσιο για την υποστήριξη της ασφάλειας και της αναθεώρησης και μεταρρύθμισης. Υπάρχει και ένα έγγραφο υπηρεσιακό εργασίας. Και υπάρχει και μέσο για τη σταθερότητα και την ειρήνη. Χρειάζεται μελέτη αντικτύπου και πάλι ένα έγγραφο εργασίας υπηρεσιακό σχετικά κυκλοφορεί. Όλα αυτά τα χαρτιά φυσικά θα τα έχετε πάρει και επίσημα στα χέρια σας ή θα τα λάβετε μόλις μεταφραστούν γιατί δεν έχουν ακόμα μεταφραστεί όλα γι' αυτό δεν έχουν διαβιβαστεί επισήμως. Τι θα λοιπόν το εξή ερώτημα που έκανε και η κυρία Χάουταλα έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με Framework Το πώς εντάσσεται αυτό σε ένα πλαίσιο. Θέλουμε να είμαστε στη δεχμή του δόρατος της ασφάλειας και άλλωστε αυτό είναι πάγια τακτική μας. Πάνω από ένα δισεκατομμύριο έχουμε δεσμεύσει για τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας. Αυτό έχει να κάνει και με τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος ή και μια σειρά άλλων νομικών δράσεων. Η ε, ε, ασφάλεια είναι ευρύτερη έννοια. Για να είναι σταθερή η κατάσταση σε μια χώρα και να επέλθει η ανάπτυξη. Αυτή η μεταρρύθμιση λοιπόν του κλάδου ασφαλείας συνδέεται με στοιχεία, ε, δηλαδή είναι με βάση δεδομένων, εμπεριστατωμένη, δεν είναι θεωρητική και τυχαία. Καταγράφονται όλα τα στοιχεία που μπορεί να περιλαμβάνονται. Λέω, είναι πραγματικά πάρα πολύ σύγχρονο έγγραφο στην αιχμή του δώρατος μαζί με τα κράτη-μέλη. Έχει συνταχθεί. Τώρα. Does indeed, um, uh, ε, επίσης, θα πρέπει σε ένα περιορισμένο βαθμό και βέβαια ε, υπό έκτακτες περιστάσεις μπορεί να συνεργαζόμαστε και με το στρατό. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορούν καμιά φορά μόνο οι στρατιωτικοί να φτάνουν σε κάποιες περιοχές για να ανταποκρίνονται στο στόχο. Το είδατε αυτό και στην ανθρωπιστική βοήθεια. Υπάρχουν περιπτώσεις που η πολιτική βοήθεια δεν φτάνει. Χρειάζονται μεταγωγές του στρατού ε, ε, για να και μεταφορές για να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια. Το ίδιο ισχύει και για την εξασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας σε μια χώρα. Δηλαδή χρησιμοποιούμε στρατιωτικούς για στόχους αναπτυξιακούς και όχι για στρατιωτικούς στόχους. Είναι ξεκάθαρο το κείμενο εδώ του μέσου. Ό,τι και να γίνει, και μόνο σε έκτακτες περιστάσεις, όταν δεν υπάρχουν άλλοι φορείς, διαθέσιμη, καταφεύγουμε στο στρατό. Όταν υπάρχει ε, σοβαρή απειλή για θεσμούς του κράτους προς τη λειτουργία τους ή όταν υπάρχει και συνένεση όλων των υπολείπων ότι μόνο μέτρα ασφαλείας μπορούν να μας εξασφαλίσουν την παροχή ε, βοήθειας. Δεν μιλάμε για τις τρέχουσες στρατιωτικές ταπάνες, ούτε για προμήθεια εξοπλισμού και πυρομαχικών. Όλα αυτά εξαιρούνται ε, και οποιαδήποτε εκπαίδευση του στρατού ε, δεν θα έχει να κάνει με το αξιόμαχο, δηλαδή δεν τους εκπαιδεύουμε ε, για να πολεμάνε, αλλά για την ανάπτυξη. Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τους. Αυτό το συμφωνήσαμε το Φεβρουάριο σε επίπεδο όσα όπου τροποποίησαμε λίγο ε, τον ορισμό της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, ODA, της κρατικής δηλαδή. Και έχουν γίνει διάφορες τέτοιες συζητήσεις. Και αυτό αφορά μόνο αυτό. Χρησιμοποιούμε το στρατό για πολιτικούς σκοπούς ή για σκοπούς αναπτυξιακούς ή όταν πρόκειται για έλεγχο των στρατιωτικών από πολιτικές δυνάμεις. Δηλαδή ε, για να μην υπάρχει βία κατά το φίλων ή για να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχει και τέτοια εκπαίδευση του στρατού που δεν είναι στρατιωτική. Και εκεί μπορεί να χρησιμοποιηθούν κονδύλια αναπτυξιακά, αλλά ποτέ για στρατιωτική δράση, επαναλαμβάνω. Γνωρίζουμε όλοι ότι εδώ εγγύζουμε τα όρια της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, ODA, ε, αλλά θα πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές, να καταλαβαίνουμε τι γίνεται σε κάθε περίσταση. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τους πόρους μας για να εγγυηθούμε την ασφάλεια, αλλιώς δεν νοείται ανάπτυξη. Κατά κάποιο τρόπο αυτό έρχεται συνέχεια στο προσκήνιο, έχουμε όλο και πιο εύθραυσες χώρες, χώρες σε πόλεμο, Κάναμε πολύ εκτεταμένες συζητήσεις με την νομική μας υπηρεσία για τους περιορισμούς που επιβάλλει η συνθήκη της Λισαβόνα και ο προπολογισμό μας. Γιατί και τα δύο έχουν να κάνουν με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη σε κάποιο βαθμό και θα πρέπει να δούμε τι θα πει και ο νομοθέτης που είναι τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμεί μια πρόταση κάναμε και προσπαθούμε να ε, διευρύνουμε κάπως τα όρια, αλλά χωρίς να τα ξεπεράσουμε. Κανείς δεν είπε να υποστηρίξουμε το στρατό, ας πούμε, για μάχημους σκοπούς. Με εξαίρεση, που δεν θέλω να σας κρύψω, που είναι η, η Αφρικανική Διευκόλυνση για την Ειρήνη, όπου χρηματοδοτούμε μέρη ε, τα αφρικανικά στατεύματα μέσω της ε, ε, Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης για την επιβολή και διατήρηση της ειρήνης στη Σομαλία. Αυτό είναι διαφορετικό όμως και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη δεν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, τον ενωσιακό. Ε, πραγματικά κινούμαστε στα όρια των προγραμμάτων, αλλά αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να δράσουμε. Και θα ήταν οτιδήποτε αντίθετο εις βάρος των στόχων μας για την ανάπτυξη. Η νομική βάση είναι στη συνθήκη της Λισαβόνας στο άρθρο για την ανάπτυξη. Και οτιδήποτε συμφωνηθεί θα μπει σε ένα τέτοιο ταμείο και θα έχει βασικό στόχο την ανάπτυξη. Αυτά μπορώ να σας πω. Δεν ξέρω, μπορεί να θέλετε προφανώς πιο επίσημη πολιτική απάντηση από τον Επίτροπο, αλλά αυτό μόνο σε απότερο στάδιο μπορεί να γίνει. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Χαότολα, θέλει να επανέλθει. Um, Νομίζω πως... Ε, είναι λίγο πράγματι ασαφής η κατάσταση σε ό,τι αφορά αυτούς τους ε, στόχους της αναπτυξιακής βοήθειας ε, και έτσι χαρμινεύσει και αυτή την τροποποίηση σε ό,τι αφορά αυτών των μηχανισμών για την συνεισφορά, για την σταθερότητα και την ειρήνη. Άρα λοιπόν το ερώτημα που θα πρέπει να θέσουμε από εκεί και μετά είναι γιατί τα κράτη-μέλη δεν αξιοποιούν τις υφιστάμενες δυνατότητες που έχουν για τη χρηματοδότηση αυτών των δραστηριοτήτων ε, που σχετίζονται με τις ενόπλες δυνάμεις. Υπάρχει το πρόγραμμα Αθήνα και υπάρχει και το known paper από από κράτη-μέλη της 15 η Απριλίου με τίτλο Food for Thought το οποίο ουσιαστικά δίνει την εντολή στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση να εφαρμόσει τα όλα όσα μα είπατε. Οπότε, σα ρωτώ, αυτό το non-paper έχει δημοσιευθεί και έχει γίνει μια δημόσια συζήτηση. Γιατί όταν έχουμε μια τόσο σημαντική ε, αλλαγή η οποία ουσιαστικά φτάνει στα όρια και ε, κατά την άποψή μου κινείται και πέραν των ε, νομικών ορίων που προβλέπονται. Και με αυτό δεν θα χαρεί σίγουρα η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η κατάσταση σχέση με αυτό το έγγραφο. Πώς δημοσιεύθηκε και ποια θέση έχουν υιοθετήσει τα κράτη-μέλη. Νέα κράτη-μέλη είπαν λοιπόν, δεν θα υπάρξουν νέα κονδύλια. Οπότε 100 εκατομμύρια ευρώ θα ληφθούν από τους μηχανισμούς της αναπτυξιακής συνεργασίας. Θεωρείτε εσείς λοιπόν από πλευρά της Επιτροπής ότι θα πρέπει να σεβαστούμε μια τέτοια απόφαση, μια τέτοια τροποποίηση. Κλάος, έχεις πολύ το λόγο. Ναι, καταρχήν θα ήθελα να πω ότι τα 100 εκατομμύρια αποτελούν μια δυνατότητα. Δηλαδή, ε, ουσιαστικά μέσω αυτής της πρότασης λέμε ότι ακόμα ε, θα πρέπει να βρούμε τα κονδύλια ε, ούτως ώστε να προσθεθούν σε αυτό το μηχανισμό για τη σταθερότητα. Σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να κάνουμε μια μεταβίβαση κονδυλίων εντός της γραμμής 4. Ε, Οπότε ε, ακόμα και σε εκείνη την περίπτωση αυτό το ζήτημα θα τίθεται πάλι προς έγκριση στο Κοινοβούλιο. Θα μπορούσαμε ένα μικρό κομμάτι των κονδυλίων της ΕΕ να επενδυθούν εκεί αλλά 100 εκατομμύρια μόνο, που αποτελεί βέβαια ένα μικρό κομμάτι. Αλλά και αυτό ακόμα δεν έχει αποφασιστεί. Αναφέρεται και αυτό ως δυνητικό σενάριο. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό το non-paper των 900 μελών, ναι, εκείνα τα κράτη-μέλη θα ήθελαν να κινηθούν ε, πολύ πιο πέρα και ε, είναι αλήθεια και το περιγράψατε. Ε, δεν γνωρίζω αν έχει δημοσιευθεί. Είναι ένα non-paper από πλευρά 9 μελών, έχει διανεμηθεί στο Συμβούλιο, αλλά δεν ξέρω ποια ακριβώς είναι το status αυτού του εγγράφου. Αυτά λοιπόν πάντως τα κράτη-μέλη θέλουν να κινηθούν ακόμα πιο μακριά γιατί με βάση τη δική τους ανάλυση οι ανάγκες ειδικότερα σε πολλές αφρικανικές χώρες οι ανάγκες λοιπόν ε, ε, ασφαλές των, των, των, των ε, είναι πολύ πιο αυξημένες και είναι απαραίτητο αυτό γιατί σε αυτή την κατάσταση αυτές οι δυνάμεις δεν είναι σε θέση να εγγυηθούν την ασφάλεια. Για παράδειγμα στην Σομαλία οι Εθνικέ Ενόπλε δυνάμει δεν είναι σε θέση να προστατεύσουν τη χώρα από την Al-Shabaab. Και υπάρχουν άλλοι ε, ε, στρατιώτε από άλλε δηλαδή αφρικανικές χώρες οι οποίε προστατεύουν τη Σομαλία από την Al-Shabaab γιατί ακριβώ η Σομαλία δεν μπορεί να το κάνει μόνη τη. οπότε αυτό είναι ένα παράδειγμα για τι προκλήσης που αντιμετωπίζουμε σε αυτό το επίπεδο. Τώρα, ω προ το ερώτημα του γιατί τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να αξιοποιήσουν άλλου υφιστάμενου μηχανισμού υπάρχουν ε, τα CFSP και Αθήνα, αλλά αυτά μπορούν να χρηματοδοτήσουν μόνο ε, ενόπλε δυνάμει ευρωπαϊκών ε, κρατών. Δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενόπλε δυνάμει αναπτυσσόμενων χώρων. Και γι' αυτό οι διάφορε στρατιωτικέ δράσει, για παράδειγμα στη Μεσόγειο ή στον Δικό Ωκεανό, γίνονται υπό την ηγεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι υπό τι ενόπλε δυνάμει των χωρών εταίρων. Άρα λοιπόν πραγματικά εδώ σε ό,τι αφορά το τους διάφορους μηχανισμούς και τα εργαλεία που διάθεσή μας, υπάρχει ένα κενό σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Άρα με βάση τα εργαλεία που έχουμε αυτή τη, σε αυτή τη φάση στη διάθεσή μας δεν μπορούμε να καλύψουμε αυτό το χρηματοδοτικό κενό ε, και μέχρι το ε, ε, επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο σε 3-4 χρόνια θα υπάρξει μια ολόκληρη συζήτηση γιατί υπάρχουν κάποια κρατημέλη που θέλουν να καλυφθεί αυτό το κενό, αλλά βέβαια είναι πολιτικό ο διάλογο και βρισκόμαστε στι απαρχέ αυτού του πολιτικού διαλόγου. Αλλά σα ξαναλέω, η εργαλειοθήκη που έχουμε αυτή τη ε, σε αυτή τη φάση, δηλαδή οι υφιστάμενοι ε, μηχανισμοί χρηματοδότησης δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε αυτό που προτείνεται με την διεύρυνση του ε, μηχανισμού χρηματοδότησης για τη σταθερότητα και την ειρήνη. Ωραία, θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε όλα αυτά, γιατί θα έχουμε προτάσεις από την Κομισιόν. Θα πρέπει μάλλον να καλέσουμε την είπατε εκπρόσωπο κάποια στιγμή να έρθει να μας εξηγήσει την πρόταση και σας ευχαριστώ ευχαριστώ Χέντι που έθιξε στο θέμα 19 διάφορα στην ημερήσια διάταξή μας Δεν μου έχει αναφέρει κανείς τίποτα για τα διάφορα. Να ευχαριστήσω τους Βερμινείς σήμερα πάντως. Τελευταία φορά που σας βλέπουμε πριν το καλοκαίρι. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για θαυμάσια δουλειά που κάνατε και δερμή ευχαριστώ την Πρόεδρο. Συνάδελφοι, όσοι δεν έρθετε στην επόμενη συνεδρίαση με την ΑΦΕ, τώρα σας εύχομαι καλό καλοκαίρι και θα τα πούμε σύντομα. Ευχαριστώ. Πέρα στη συνεδρία σα. Α, 2Q2 για την συνεδρίαση με την ΑΦΕΤ έχει καθυστερήσει 10 λεπτά. 10, συγγνώμη, 5 ε, και 10. 5 και 10 αρχίζει, σε 10 λεπτά δηλαδή.